We Μπορούμε να ξαναρχίσουμε τη δουλειά μας αν είστε έτοιμοι αγαπητοί συνάδελφοι. Okay. So welcome back. Happy to start again. Καλώς ήρθατε και πάλι χαίρομαι που είμαι εδώ κοντά σας να ξαναρχίσουμε τη δουλειά μας μετά τις θερινές διακοπές. Ένα-δύο σοβαρά θέματα συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού με την Κόσια. Καταρχάς, σε διάταξη. Αντιρρήσεις δεν βλέπω. Ανακοινώσεις δεν έχω. Ίσως με τους συντονιστές να οργανωθούμε για να, κάνουμε, να πάρουμε αποφάσεις και έτσι θα έχουμε αύριο ανακοινώσεις μάλλον. Έγκριση πρακτικών της 10 η Ιουλίου της πρώτης συνεδρίασής μας. Αντιρρήσεις δεν βλέπω, Εγκρινώνται λοιπόν τα πρακτικά και προχωρώ κατευθείαν στο σημείο 5 Τη ημερήσια δέταξη μα πάει έω τι 10.30 γιατί εσεί μετά θα πρέπει να αποχωρήσετε στι 10.30. Χαίρομαι λοιπόν που έχω εδώ φιλοξενούμενο τον κύριο Χολολάη με ένα θέμα καυτό την Κόρσια και πώς αντιλαμβανόμαστε το θέμα αυτό ή το Κόρσια που συζητούμε και με την ΙΚΑΟ ε, σε σχέση με ε, την εξασφάλιση ενός παγκόσμιου διεθνούς οργανισμού ή μηχανισμού που θα επιτρέψει τον περιορισμό και την απόσβαση των ε, ανθρακούχων εκπομπών και τον κίνδυνο που διατρέχει να αποτύχει. Αυτό περιμένουμε λοιπόν εμείς σήμερα ελπίζουμε απαντήσεις και πάνω απ' όλα ελπίζουμε να μας διαβεβαιώσετε πως δεν υπάρχει ο κίνδυνος. Αλλά μάλλον δεν θα τα ακούσουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το κύριο κίνητρο που μας οδηγεί στη, στη διοργάνωση αυτής της ε, ακρόασης. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και σας δίνω 10 με 15 λεπτά για να, ξεκινήσετε για να κάνετε την ε, παρουσίαση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, είπατε κι εσείς ότι είναι καυτό το θέμα ελπίζω και το καλοκαίρι σας να ήταν τουλάχιστον ζεστό και ευχάριστο. Α, κάπου κάπου. Εκεί που ήμουν εγώ έβρεχε συνέχεια ή σχεδόν. Και έτσι γυρνάω με χαρά. Αν και φαντάζομαι όλοι επιστρέφουμε με χαρά. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Και ξεκινώντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Κονφέν, κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση που είχε απευθυνθεί αρχικά στην Επίτροπο Μπούρτς, η οποία όμως δεν μπόρεσε δυστυχώς να ε, έρθει και έτσι με παρακάλεσε να την αντικαταστήσω. Με χαρά λοιπόν ε, θα σας ενημερώσω για την επερχόμενη σύνοδο της 40ης ΙΚΑΟ και την Κόρσια. Το πρόγραμμα λοιπόν περιορισμού και απόσβεση των εκπομπών του άνθρακα στις διεθνείς αερομεταφορές. Ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με τον περιορισμό του περιβαλλοντικού ίχνους και της περιεκτικότητας σε άνθρακα, των εκπομπών άνθρακα των μεταφορών που έχουν καταστεί άλλωστε και μεγάλη προτεραιότητα της Προέδρου, της ε, στη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίας Φόντερ Λάιεν. Έχουμε ένα 2% σε ποσοστά εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου στην αεροπορία. Έχουμε ένα σημαντικό περιορισμό τα τελευταία χρόνια, μείον 24% από το 2004 στο 2017 του μέσου, της μέσης ποσότητας ε, εκπομπών, μάλλον χρήσης ε, καυσίμων, αλλά χρειάζεται ακόμη περισσότερες ε, προσπάθειες. Έτσι λοιπόν με την παρουσίαση των πολιτικών ε, κατευθυντηρίων γραμμών για την προσοχή επιτροπή τον Ιούλιο, η κυρία Φόντερ Λάιεν επεσήμανε ότι η επιτροπή θα είναι φιλόδοξη περισσότερο προς τον περιορισμό και την επίτευξη του στόχου της ουδετερότητας της κλιματικής στο 2050 περισσότερο δηλαδή φιλόδοξη από ότι το έχει οριστεί για ένα περιορισμό έως το 2030 στο 40% των εκπομπών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει και η αεροπορία και η πολιτική φυσικά να ε, περιορίσει τις εκπομπές της, να κάνει προσπάθειες κοινέ με τον τομέα των μεταφορών και έτσι μιλούμε για ένα παγκόσμιο βεληνικού σχέδιο, το Κόρσια, που έχει κρίσιμη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου να πω ότι το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Κόρσια γενικότερα και που εκδηλώνεται από πλευρά κυρίω των Επιτροπών, αλλά και γενικότερα και που εκδηλώνεται κυρίω από πλευρά των Επιτροπών ΕΝΒΙ και ΤΡΑΝΕ, το θεωρούμε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Έχουμε την 40η Γενική Συνέλευση τη ΣΥΚΑΟ στο Μόντρεαλ στο τέλο του μήνα με μια ε, κατεύθυνση που θα δοθεί όπως κάθε φορά στις ε, ανατριετή αυτές συνεδριάσεις των εκπροσώπων των κρατών μελών της ΙΚΑΟ και που θα ορίσουν βέβαια με τον τρόπο αυτό την πολιτική και τις τάσεις για τα επόμενα τρία χρόνια με ε, την ελπίδα για μας να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι εκπομπές από την αεροπορία. Αυτό σημαίνει και για να καταπολεμήσουμε βεβαίως την κλιματική αλλαγή, να έχουμε μια ουδέτερη ανάπτυξη ως προς τις εκπομπές άνθρακα από το 2020 και μετά. Για το 2016 εξασφαλίστηκε μια ιστορική συμφωνία ώστε να τεχθεί ένα πρώτο στην ιστορία σχέδιο περιορισμού των εκπομπών με ιδιαίτερα ενεργή, ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπόρεσε να πείσει τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΚΑΟ και ε, ιδιαίτερη υποστήριξη από αρκετούς ευρωβουλευτές μεταξύ των οποίων και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής σας κύριος Σίκχαουτ που μπόρεσαν υποστήριζοντάς μας να εξασφαλίσουν λύσεις και αποφάσεις που δεν είχαν φανεί εύκολες στην αρχή. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα μηχανισμό, το Corsia ή την Corsia, που ζητεί από τις ε, αερογραμμές να εξουδετερώσουν την αύξηση ε, των εκπομπών σε διοξίδιο του άνθρακα από, σε σχέση με το επίπεδο που θα έχουν φτάσει το 2020 και μετά με εθελοντικό, εθελοντική συμμετοχή από το 2021 στο 2026 και υποχρεωτική από το 2027 με παρακολούθηση, αναφορές, επαλήθευση και εξασφάλιση αξιόπιστων δεδομένων μπορούμε να έχουμε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Πέρασαν λοιπόν τρία χρόνια από αυτή την ε, Γενική Συνέλευση. Έχουν εγκριθεί εντωμεταξύ οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του σχεδίου και έχουμε μέσα στη διαδικασία αυτή αγωνιστεί και έχουμε την ανάγκη να αγωνιστούμε για ένα φιλόδοξο σχέδιο. Ε, έχουμε απέναντί μας αντιμέτωπα κράτη τα οποία δεν θέλουν να έχει τόσο αυστηρές ε, προδιαγραφές και περιγραφές στο σχέδιο Κόρσια. 81 είναι τα κράτη με 76% των δραστηριοτήτων στην διεθνή αεροπορία που έχουν δεχθεί να συμμετάσχουν εθελοντικά στην πρώτη πιλωτική φάση από το 2021 και μετά, πράγμα το οποίο θεωρούμε μεγάλη επιτυχία. Το Κόρσια μπορεί να είναι ίσως όχι ε, ε, θα είναι το καλύτερο και αν, όχι και το μόνο εργαλείο που θα έχουμε για τον περιορισμό των κλιματικών συνεπειών της αεροπορίας και άρα την τήρηση των συμφωνιών του Παρισιού στο τομέα της αεροπορίας. Γιατί το ETS και μόνο του με όλες τις φιλοδοξίες ε, που έχει και είναι υψηλές δεν θα επαρκέσει για να αντιμετωπίσει επαρκώς το πρόβλημα των εκπομπών από τις παγκόσμιες αεροπορικές μεταφορές και έτσι θα πρέπει και ε, όλα τα κράτη της ΙΚΑΟ να συμμετάσχουν στο Κόρσια, αλλά και να επιταχυνθεί ενδεχομένως το βήμα που θα ακολουθήσει η αεροπορία στην ενσωμάτωση του Κόρσια σε όλο τον κόσμο για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε πολύ δύσκολες αισθήσει πραγματοποίηση, γιατί υπήρξαν αμφισβητήσει προς την αποκλειστικότητα του Κόρσια και κατά πόσο είναι το μόνο εργαλείο που στηρίζεται στην αγορά για τον περιορισμό των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα ε, στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Ιούνιο φέτος. Εν τω μεταξύ έχουμε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ε, στις οποίες τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν κρατήσουν εκείνων που ήθελαν να διατηρηθεί μια αναφορά στο αποκλειστικότητα ως όρο για το Κόρσια. Ε, και έτσι έχουμε μία πρόταση η οποία θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια ε, θέση για το Κόρσιο και παραπέμπω στο σχετικό κείμενο που θα αποτρέπει την ε, εμβαλωματική λύση επαναλαμβανομένων ή επικαλυπτωμένων σχεδίων και προγραμμάτων σε παιδοκρατικό ή περιφερειακό, έτσι ώστε διεθνείς εκπομπές οι εκπομπές μάλλον του άνθρακα της Διεθνούς Αεροπορίας να καταγράφονται μόνο άπαξ. Και αυτή ήταν η προσπάθεια προς την οποία τίνουμε. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε την επόμενη χρονιά να έχουμε μια έκθεση υπεπραγμένων που θα είναι και σύμφωνη με το ETS. Το Συμβούλιο Συνομοθέτης μαζί με το Συμβούλιο θα πρέπει βάσει αυτής της εκθέσεως να αποφασίσουν πώς η Κόρσια θα ενσωματωθεί στην οδηγία για το ETS, την φυστάμενη οδηγία. Θα προσπαθήσουμε ταυτόχρονα και να πείσουμε τους ε, εταίρους τρίτα κράτη ε, πως είμαστε αποφασισμένοι το Κόρσια να το υλοποιήσουμε πλήρως και σύμφωνα με την οδηγία ETS ε και με τις γενικότερες περιβαλλοντικές φιλοδοξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους όρους λειτουργίας της αγοράς των ανταλλαγών εκπομπών. Έτσι λοιπόν, ο όρος περί αποκλειστικότητα θα κριθεί σήμερα από την Επιτροπή σε σχέση με την ορολογία που θα χρησιμοποιηθεί στην Γενική Συνέλευση ε, ώστε να εξασφαλιστεί μια λύση με ένα κείμενο της Επιτροπής το οποίο θα έρθει στη συνέχεια πει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να είναι σύμφωνο με τις δεσμεύσεις μας. Διατηρείται η αυτονομία της ε, Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Λήψη Αποφάσεων, η Σύμβαση του Σικάγο επιτρέπει, αναγνωρίζει τη δυνατότητα σε ένα κράτος μέλος αυτόνομα να λαμβάνει αποφάσεις εφόσον δεν διαταράσσουν τις ε, διεθνείς συμφωνίες και άρα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει αποφάσεις με βάση και τις συμφωνίες των Παρισίων στις διεθνείς διαπραγματεύσεις ε, πάντοτε επιδιώκουμε να διατηρούμε την ε, αυτονομία αποφάσεων ώστε να ορίζουμε υψηλότερα επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και θα ήθελα να αναφερθώ κλείνοντας κυρίες και κύριοι σε, σε μια ακόμη σειρά ε, μέτρων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να αναλάβει σε σχέση με την ε, προστασία του περιβάλλοντος. Ναι, με, ξέρω ότι με καλέσατε για να σας μιλήσω για, την, το κόρση, αλλά είναι μόνο ένα εργαλείο ε, περιορισμού των εκπομπών της αεροπορίας. Υπάρχουν λοιπόν μηχανισμοί αγοράς, το ETS, ε η Κόρσια, που βελτιώνουν τις συνθήκες των ευρωπαϊκών εθέρων και με βάση το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εθέρες με 2,6 δισεκατομμύρια εκπομπών που έχουν εξοικονομηθεί από το 2014 και που θα μπορούσαν ακόμη περισσότερο να εξοικονομηθούν εάν δεν είχαμε την παρεμπόδιση από πλευρά ορισμένων κρατών μελών στο Συμβούλιο για λήψη δράσεως. Ε, προχωρούμε και στην έρευνα, την ανάπτυξη, την ε, χρήση τεχνολογίας για βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών και στην παραγωγή κατασκευή αεροσκαφών ε, μέσα από το πρόγραμμα Καθαρή Ουρανή, τεχνολογία ε, που αναμένεται το 2025 με 27 να είναι έτοιμη, 75% ε, του στόλου αεροσκαφών που έχουμε αυτή τη στιγμή αναμένεται στο 2050 να έχει υιοθετήσει και ενσωματώσει καθαρές τεχνολογίες. Καύσιμα επίσης, καύσιμα καθαρά και αηφόρου χρήσεως ε, ε, πρέπει να είναι ένας επόμενος στόχος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα 0,05% αλλά θέλουμε να δώσουμε κίνητρα με ένα νομικό πλαίσιο που θα ενισχύει και θα υποστηρίξει τις επενδύσεις με στόχο τελικά τον περιορισμό της χρήσης της κυροζήνης και την εξασφάλιση καθαρότερων καυσίμων. Αυτή τη στιγμή βεβαίως που βρισκόμαστε σε μια φάση αλλαγής μεταξύ ε, Αλλαγή σε επίπεδο επιτροπής επιτρόπων ε, δεν είμαι σε θέση εγώ να αναλάβω ε, δεσμεύσει ή να τοποθετηθώ πιο συγκεκριμένα στο θέμα αυτό. Πάντως τα μέτρα θα έχουν να κάνουν και με την ενίσχυση των μηχανισμών της αγοράς. Η Ευρώπη θα μπορέσει στην συνέλευση της ΙΚΑΟ να επιμείνει για την ενίσχυση των επιπέδων φιλοδοξίας περιορισμού, δηλαδή των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα από το 2020 και μετά σε όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα προτινόμενα μέτρα, τεχνολογία όμως και ε, πρόοδο σε συνεργασία με, την σχετική, με το σχετικό βιομηχανικό κλάδο θα είναι κλειδιά στον περιορισμό αυτών των εκπομπών με στόχο την εξασφάλιση ωφελών ε, και για το περιβάλλον μέσα από την αεροπορία και αυτό βέβαια είναι αναμονή περαιτέρω διεθνών συμφωνιών, δεσμεύσεων και αποφάσεων. Αυτά πρόεδρε εντάχει και σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πολύ καλά τηρήσατε το χρόνο σας. Όσον αφορά την ουσία, ε, θα δούμε με τους συντονιστές μαζί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τις ερωτήσεις ε, των συντονιστών. Δύο λεπτά ο καθένας και σας παρακαλώ να παραμείνετε εντός του χρόνου που σας δίνω. Ας ξεκινήσουμε από το ΕΛΚ και τον Πέτερ Λίζε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντή. Δύο τεράστια προβλήματα υπάρχουν όσον αφορά το Κόρσια. Η ΙΚΑΟ που ανέπτυξε το Κόρσια είναι όργανο των Ηνωμένων Εθνών ε, και παραθέτω τα λόγια του Αντώνιο Κουτιέρες που ζητάει από όλα τα κράτη-μέλη από όλους τους φορείς ε, της οικονομίας να παρουσιάσουν ε, φέτος τον Σεπτέμβριο σχέδια ώστε μέχρι το 2030 να μειώσουν κατά 45% τα 100 της εκπομπές ε, και μέχρι το 2050 να είναι ουδέτεροι ως προς το κλίμα. Αυτά ζητάει ο Γενικός Γραμματέας ε, των Ηνωμένων Εθνών ε, Αντώνιο Γκουτιέρες, αλλά θα έπρεπε να ξεκινήσει από τον δικό του οργανισμό, διότι η ΚΑΟ, για να το πω χοντρά, είναι χειρότερη από τον Πολσονάρο και τον Τραμπ, διότι ο τομέας των αερομεταφορών είναι αυτός που απέχει περισσότερο από τον στόχο που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Οι εκπομπές αυξάνονται σε όλο τον κόσμο, δεν μειώνονται και ε, το σύστημα Κόρσια δεν υποχρεώνει τις αερομεταφορές να μειώσουν τις εκπομπές και δεν θα λειτουργήσει καν ο περιορισμός της αύξησης, διότι δεν ε, λειτουργεί το ε, σύστημα αντιστάθμισης, διότι είναι γεμάτο παραθυράκια. Είναι δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ζητάει ο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Και ε, είμαι λίγο απογοητευμένος που ο Γενικός Διευθυντής δεν το ε, κατέκρινε αυτό. Επίσης, έχουμε αποφασίσει οι αερομεταφορές να συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, αλλά είναι πολύ ε, χαμηλότερες οι, οι φιλοδοξίες μας στο θέμα αυτό ε, και αναρωτιέμαι πώς θα εξηγήσω σε κάποιον εργάτη της βιομηχανίας Χάλιβα ότι δεν είμαστε πιο αυστηροί. Κάποιοι ζητάνε περισσότερα και στις αερομεταφορές... Ε, κλείνω, Πρόεδρε. Κλείνω. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το εκφράσει αυτό με πολύ πιο σαφή λόγια από ό,τι ακούσαμε σήμερα από τον Γενικό Διευθυντή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για τον ε, περιορισμό του χρόνου. SND. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευκαιρία αυτή να συνομιλήσουμε μαζί σας. Για το S&D δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αντιμετώπιση των εκπομπών ε, θα πρέπει να γίνει από το σύνολο της κοινωνίας και η ιδέα του Κορσία δεν είναι άσχημη, είναι να έχουμε ένα, μια, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα, μια παγκόσμια λύση για ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Υπάρχουν ε, όμως ε, σημαντικά ελαττώματα στην πρόταση για το Κοινοβούλιο έχει στο παρελθόν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ακεραιότητα και το νόημα του συστήματος όπως για παράδειγμα την ε, αντιστάθμιση μετά το 2020 και επίσης το Κορσία ε, επιτρέπει το καθαρό πετρέλαιο, ε, το οποίο είναι εξωφρενικό. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με αυτό το, καθαρό πετρέλαιο ως εναλλακτικό καύσιμο για το Κορσία ή τι κάνει για να εξαλείψει αυτό το παραθυράκι. Και επιπλέον το σχέδιο κειμένου αναφέρει ότι το Κορσία είναι το μόνο παγκόσμιο μέτρο για την αντιμετώπιση των ε, εκπομπών ε, στις αερομεταφορές ε, και αποκλείει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει για να βεβαιωθεί ότι το Κορσία δεν θα υπονομεύσει το δικό μας σύστημα εμπορίας εκπομπών και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την αντίδραση των άλλων χωρών. Και τέλος, στην Ευρώπη δεν κάνουμε αρκετά για να μειώσουμε τις δικές μας εκπομπές. Η δική σας μελέτη για την φορολογία και τις εκπομπές δείχνει ότι υποφορολογούνται οι αεροπορικές εταιρείες. Ε, πιστεύετε λοιπόν ότι είναι αιτιολογημένη αυτή η στάση ή θα υποβάλλετε συγκεκριμένες προτάσεις για να εξαλείψετε αυτό το παραθυράκι που υπάρχει όσον αφορά τις εκπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ. Από το Renew, ο Νίλ Στόρβαλς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Γενικέ Διευθυντά που βρίσκεστε εδώ πέρα, αν και μπορεί να είναι κάπως αμήχανη η συζήτηση αυτή για σας. Όπως ήδη ακούσατε, η βασική μας επιφύλαξη είναι ότι η διατύπωση στο Κορσία και στο ψήφισμα υπονομεύει την ακαιρεότητα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα επιμείνει όλα τα κράτη-μέλη είτε να απορρίψουν την πρόταση ή αν δεν το καταφέρει αυτό να υποβάλουν επιφυλάξεις ε, σε σχέση με την πρόταση και τι συγκεκριμένες συνέπειες για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υπάρξουν από την ε, διατύπωση. Όπως είπε και η κυρία Γκούτελαντ, μας ανησυχεί η φράση ότι είναι το μόνο παγκόσμιο μέτρο που βασίζεται στην αγορά. Πολύ θα ήθελα να μας δώσετε όσο γίνεται πιο σαφείς απαντήσεις στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τους πράσινους, ο Μπάς Έιχουτ. Στα δεξιά σας ε, κάθομαι. Ε, καλημέρα και σας ευχαριστώ κύριε Χολολαή για την εισαγωγή σας. Νομίζω ότι ήδη θα ακούσατε από τους συναδέλφους μου ότι η έλλειψη εξελίξεων στην ΙΚΑΟ θα έλεγα μας ανησυχούν επίσης μας ανησυχεί η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί τόσο έντονα μια παγκόσμια λύση και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτή είναι η προτιμητέα λύση, διότι ε, καλύτερο θα είναι όλοι να κινηθούμε. Ωστόσο, η πρόοδος ε, εντός της ΙΚΑΟ ήταν τόσο ε, ελάχιστη όσον αφορά τις προτάσεις αποφάσεων που ήρθε η ώρα να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ΙΚΑΟ ότι ε, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ε, τα θέματα των εκπομπών στον τομέα αερομεταφορών, ακόμα και αν η ΙΚΑΟ δεν κάνει τίποτα. Ε, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να απορρίψουμε την διατύπωση ω έχει το ότι το Κόρσια δηλαδή θα πρέπει να είναι το μόνο σύστημα και αν υιοθετηθεί θα πρέπει να στείλουμε σαφές μήνυμα, να υποβάλουμε επιφύλαξη και δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο ακόμα. Ε, γι' αυτό μήπως μπορείτε να είστε πιο σαφείς στο θέμα αυτό. Και επίσης ε, όσον αφορά τη διατύπωση, λέμε ότι το αν ε, θα συμμετάσχουμε εξαρτάται από την περιβαλλοντική ακαιρεότητα των κανόνων αυτό το λέει η νομοθεσία που αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα ε, Εμπορίας Εκπομπών. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, πιστεύετε ότι οι κανόνες για την αντιστάθμιση ε, είναι περιβαλλοντικά ακέραιοι. Δεν το πιστεύω, ούτε νομίζω ότι πολλοί άλλοι το πιστεύουν αυτό. Μπορείτε παρακαλώ να είστε σαφείς όσον αφορά το θέμα αυτό. Και το ίδιο ισχύει για τα εναλλακτικά καύσιμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο σαφή διατύπωση και πιο σαφείς θέσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στην ε, ΙΚΑΟ και θα ήθελα να ακούσω πιο σαφή λόγια από τον κύριο Χολολάη. Από το ID Σίλβια Σαρντόνε. Not... Από ό,τι φαίνεται δεν είναι παρούσα. Υπάρχει κάποιος άλλος από το ID? Από το ECR, ο κύριος Βόντρα. Uh, thank Ευχαριστώ πολύ. Τρία σημεία. Καταρχήν, πιστεύω πως είναι παγκόσμιο το πρόβλημα με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και θα απαιτηθεί μια παγκόσμια αντιμετώπιση. Ε, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα η ύπαρξη της Κόρσια ή του Κόρσια και πιστεύω πως θα πρέπει να σπρώξουμε έτσι ώστε να καταφάρει περισσότερα. Το πιο ουσιαστικό είναι πως τουλάχιστον υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ο ΙΚΑΟ είναι ο μόνος οργανισμός παγκοσμίως που προσπαθεί να βρει κάποια λύση. Δεύτερον, Έχουμε κάποιο τρόπο να επηρεάσουμε τα πράγματα εάν δεν μας ικανοποιήσει ο βαθμός πρόοδου σε επίπεδο ΙΚΑΟ πόση δύναμη έχουμε στα χέρια μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να τους πιέσουμε για να προχωρήσουν παραπάνω. Η απέτηση είναι μια παγκόσμια λύση και δεν μπορεί να προσφέρουμε κάτι μόνο τοπικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τρίτο είναι πως έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην ε, απελευθέρωση της, ε, των αεροπορικών μεταφορών τα τελευταία χρόνια. Και λόγω ακριβώς αυτής της απελευθέρωσης όλοι έχουν πρόσβαση στην Ευρώπη. Πριν από 20 χρόνια ταξίδευαν αεροπορικά μόνο οι πλούσιοι, το θυμάμαι. Αν λοιπόν προωθούμε αυτό το ζήτημα ακόμα πιο πολύ, τότε οι επιπτώσεις τοπικά στην Ευρώπη θα είναι οι αερομεταφορές πια ε, να είναι προσβάσιμες μόνο από ανθρώπους πλούσιους όπως εμείς. Τι κάνουμε λοιπόν έτσι ώστε να επιτρέψουμε αυτός ο είδος μεταφορών να είναι ε, προσιτές και για τον απλό άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σίλβια Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς κύριε Γενική Διευθυντά για την παρέμβασή σας και πρέπει να σας πω πως θα συνταχθώ με πάρα πολλά από τα λεγόμενα των ε, συναδέλφων. Χρειαζόμαστε ε, ένα επαρκές επίπεδο φιλοδοξίας και παρόλα τα όσα έχουν ακουστεί και παρόλες τις φιλοδοξίες ε, προσπάθειες που έχουν γίνει το σύστημα μοιάζει να είναι μία απλή προσπάθεια ε, φτιασιδώματος του προβλήματος. Ο στον κλάδο αυτό είναι πολύ δύσκολο να μειώσει κανεί τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Είναι παγκόσμιο κλάδο, αλλά καλό θα ήταν να είχαμε ένα παγκόσμιο σύστημα μειώσεων. Επαναλαμβάνω όμω, κάτι τέτοιο θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Τι θα συμβεί, για παράδειγμα, αν κάποια χώρα θέσει πάρα πολύ φιλόδοξους στόχους έτσι ώστε να χρησιμοποιεί βιοκεροσύνη, ε, και να ταξιδεύουν τα αεροπλάνα μόνο με τις δεξαμενές γεμάτες για να μειωθεί η χορύπανση. Μπορεί αυτό να ε, εφαρμοστεί ως μεμονωμένο κρατικό μέτρο. Όχι, θα είναι αρνητικές οι επιπτώσεις. Άρα λοιπόν παγκόσμιες λύσεις. Τώρα, για το σύστημα αντιστάθμισης εκπομπών, αυτές οι χαλαρές ε, πιστώσεις οι οποίες αποκτούνται θεωρητικά για να ελαφρύνουν τη βλάβη από τις επιπτώσεις, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πως όντως μειώνουν το πρόβλημα. Γιατί μήπως τελικά αυτές δεν είναι αντισταθμιστικές πράξεις, αλλά ε, νομοθεσία που έτσι κι αλλιώς επρόκειτο να εφαρμοστεί. Γιατί δεν μπορεί αλλα νομοθεσια ένας κλάδος να αντισταθμίζει τις εκπομπές του άλλου. Νομίζω ότι αυτό θα μας οδηγήσει σε παράδοξες καταστάσεις. Επίσης έχουμε και άλλα είδη μεταφορών και συγκοινωνιών που είναι εξίσου ε, ρηπογόνα. Οπότε η φορολόγηση της ε, κεροσύνης ως καυσίμου, ναι, αποτελεί μια λύση, αλλά όχι τη μόνη. Γιατί δεν μπορούμε κάποιος ο οποίος ταξιδεύει με το αυτοκίνητό του να πληρώνει ε, φόρο στη, στη βενζίνη που καταναλώνει και αντίστοιχα να μην επιβαρύνεται η κεροσύνη με ένα ε, τέτοιο αντίστοιχο φόρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έγιναν λοιπόν οι πρώτες ερωτήσεις που ήταν πολύ συγκεκριμένες κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου και ξέρω πως αυτή τη στιγμή τρέχει μια διαδικασία, ε, επηρεάζεται από κάποιους νομικούς περιορισμούς, αλλά ίσως ε, καλό θα ήταν μέσω αυτής της ε, συνάντησης που έχουμε να ξεκαθαρίσουμε την θέση της δικής σας, θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους συντονιστές για τις ερωτήσεις και τα σχόλια που έκαναν. Πολύ σωστά είπατε κι εσείς δεν ήταν εύκολες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Το σχέδιο Κόρσια δεν είναι τέλειο. Αυτό είναι σαφές. Παρ' όλα αυτά είναι το μοναδικό παγκόσμιο εμβέλειας σχέδιο. Και μάλιστα χρειαστήκαμε πάρα πολύ χρόνο για να φτάσουμε εκεί που είμαστε σήμερα. Παραθυράκια υπάρχουν πάρα πολλά. Στοιχεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης Βεβαίω και υπάρχουν. Ξέρετε όμως πως οι διεθνεί ε, διαπραγματεύσει ε, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις πολλών διαφορετικών ε, περιοχών. Και όπως είπα και στα εισαγωγικά μου σχόλια, η Ευρώπη έδειξε πυγμή, επιχειρηματολόγησε υπέρ της μέγιστης φιλοδοξίας που είναι αδύνατη αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχει την πλειοψηφία στα χέρια της. Και το πιο σημαντικό είναι να βρούμε ποια θα είναι αυτή η πλειοψηφία που θα μας επιτρέψει ε, μέσα αυτών των 81 χωρών, που είναι το 76% των εκπομπών, να θέσουμε σε εφαρμογή το Κόρσια. Αυτό θα αποτελέσει τη σωστή απόκριση σε μια παγκόσμια πρόκληση. Και βεβαίως θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξη. Και βεβαίως προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι πιο φιλόδοξο εδώ. Βρισκόμαστε σήμερα και είναι πολύ σημαντικό ε, το Κόρσια να ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Ήδη κάπου έχει ξεκινήσει γιατί υπάρχουν κάποια ε, κράτη τα οποία ενδεχομένως δημιουργούν πολλές εκπομπές και θα γίνουν τμήματα του Κόρσια. Ε, πρέπει να τους πείσουμε έτσι ώστε σε παγκόσμιο επίπεδο να έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Πιέζουμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε. Δεν νομίζω ότι αυτό το αμφισβητεί κανείς, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως το σχήμα αυτό δεν είναι τέλειο. Είναι όμως το μοναδικό που αυτή τη στιγμή είναι στη θέση του και είναι παγκόσμιο. Το βασικό θέμα συζήτησης σήμερα είναι η αποκλειστικότητα. Και χαίρομαι που και ο ίδιος ο Πρόεδρος υπογράμμισε πως αντιμετωπίζουν νομικές, ε, νομικούς περιορισμούς επειδή ακριβώς τρέχουν κάποιες διαπραγματεύσεις και δεν μπορώ να μιλήσω τελείως ανοιχτά. Προσπάθησα όμως στα εισαγωγικά μου σχόλια να στο δυνατόν πιο σαφής Και εδώ θα επαναλάβω ποια είναι η κατάσταση. Η απόφαση της ε, συνέλευσης του ΙΚΑΟ δεν είναι νομικά δεσμευτική ε, για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά η ευρεία ερμηνεία της ρήτρα αποκλειστικότητας είναι πως οποιοδήποτε μέτρο που εφαρμόζεται ε, στην διεθνή αεροπλοεία θα πρέπει να εφαρμόσει το Κόρσια χωρίς να ανοίγει χώρο για οποιοδήποτε άλλο μέτρο, καθεστώς ή φορολογική υποχρέωση παρόμοια εμβέλειας παρά μόνο όσων μετα... Ε, εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο. Αυτό δεν έχει να κάνει με την αυτονομία των κρατών να νομοθετήσουν, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω πως εδώ εμείς δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε και καλούμε μάλιστα ε, τα κράτη-μέλη να δράσουν στη συνέλευση του ΙΚΑΟ με έναν τρόπο που δεν θα ψαλιδίσει τη δυνατότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω Κόρσια. Και βεβαίως δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Επιτροποί σήμερα και αν θα εγκρίνουν ή όχι, αλλά ε, έχουμε προτείνει να υπάρχει αυτή η αποκλειστική ε, ρήτρα ως διατύπωση στα κείμενα της ε, συνέλευσης και θα σας σταλεί και σας για ε, λόγους διαβούλευσης. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται με έναν τρόπο που θα στραφεί εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εφαρμογή του Κόρσια αυτό το κείμενο. Γιατί διαφορετικά δεν θα είμαστε σε θέση να επιδιώξουμε ένα φιλόδοξο, μια φιλόδοξη πολιτική για τις αεροπορικές μεταφορές εδώ Κάτι το οποίο επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αντίστοιχη διατύπωση θα υποβάλουμε τώρα, θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη, αλλά νομίζω πως πιο ανοιχτά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω, χωρίς να παραβιάζω τους περιορισμούς ε, που μου επιβάλλονται. Εσείς βέβαια μπορείτε να καταλήξετε στα δικά σας συμπεράσματα. Ξέρω πως οι συντονιστές ε, εκφράστηκαν, ε, τους άκουσα πολύ προσεκτικά, ξέρω ποια είναι η θέση της Επιτροπής σας και ξέρω και εσείς πώς αισθάνεστε για το θέμα αυτό της αποκλειστικότητας. Έχουμε κάποια ακόμα σημεία τι γίνεται με τα καύσιμα. Το σχολίασαν και οι σοσιαλιστές. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω πως στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα χαμηλής περιεκτικότητας σε του άνθρακα καύσιμα, τα οποία αυτή τη στιγμή ε, δεν έχουν συμφωνηθεί, αλλά θα ε, συζητηθούν και θα ψηφιστούν στον ΙΚΑΟ, θα σέβονται τις ε, κατάλληλες προϋποθέσεις. Η συζήτηση αυτή, και θα σας το πω, δεν θα γίνει στην τρέχουσα συνέλευση, αλλά ε, τα επόμενα τρία χρόνια αλλά εν πάση περιπτώσει για τα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα ορυκτά καύσιμα για την μετά το κόρσια, και μάλιστα για, τους, για το μηχανισμό αντιστάθμισης εκπομπών κόρσια είναι ένα θέμα το οποίο είναι στο τραπέζι και ε, το συζητάμε στις διαπραγματεύσεις. Όμως δεν υπάρχει πρόβλημα μετακύλησης στις συζητήσεις για τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, γιατί δεν θεωρούνται βιώσιμα τα, βιώ... τα ορυκτά καύσιμα, οπότε εκεί δεν θα αντιμετωπιστεί πρόβλημα. Επαναλαμβάνω όμως, οι διαπραγματεύσεις ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Επίσης, για το μηχανισμό αντιστάθμισης και το όσα είπε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Οι κανόνες αυτοί, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους Εμπειρογνώμονες, είναι αρκετά καλοί. Το Τεχνικό Συμβουλευτικό Όργανο για την εφαρμογή και την αποδοχή των Αντιστασμητικών μέτρων αποτελείται από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες εμείς αυτό που κάνουμε είναι να παρακολουθούμε στενά τη δράση τους και στον πρώτο κατάλογο ε, των αντισταθμιστικών μέτρων ε, τον περιμένουμε τέλη του 19 μέσα στο 20 και ξεκάθαρα έχουμε περιγράψει τη θέση μας πάντα λέγοντας πως επιθυμούμε τα μέτρα αυτά τα αντισταθμιστικά να είναι ποιοτικά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταφέρουμε. Το δικό σας μήνυμα είναι σαφές, αλλά και η δική μας θέση, κατά τη γνώμη μου, έχει δείξει απόλυτη συνοχή. Και το τελικό αποτέλεσμα δεν εξαρτάται μόνο από την Ευρώπη, αλλά όπως είπα και κατά τη διάρκεια πολλών από τις συζητήσεις που είχαμε, χάρη στις ευρωπαϊκές συμφωνίες και συμβάσεις, καταφέραμε να προχωρήσουμε προς πιο φιλόδοξα αποτελέσματα. Να πω δύο λόγια και για τη φορολογία, ε, τον, τη φορολόγηση των καυσίμων ως επιπλέον μέτρο. Πάλι με φέρνετε σε δύσκολη θέση γιατί δεν μπορώ να προδικάσω το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη νέα της σύνθεση. Αυτό αποτελεί ε, θέμα των επόμενων επιτρόπων και εδώ ως αξιωματούχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είμαι σε θέση να προδικάσω τις αποφάσεις τους. Σίγουρα όμως ακούσατε τα όσα δήλωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ε, μόλις εκλεγήσα πρόεδρος και τα σχόλιά της για τη μάχη για την καταπολέμηση του προβλήματος της αλλαγής του κλίματος, και τα παραδοτέα και τα μέτρα τα οποία έχει κατά νου. Τρέχουν δε κάποιες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε σε αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία όταν ε, βρίσκεται στο τραπέζι θέμα εξαιρέσεων από την ε, οδηγία για την φορολογία των καυσίμων και νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος που θα μας επιτρέπει να εξετάσουμε διάφορες εναλλακτικές και να σημειώσουμε πρόοδο. Τώρα θα ήταν δίκαιο σε αυτή τη φάση να πω και το εξή. Όλα τα εναλλακτικά σενάρια είναι πάνω στο τραπέζι. Πρέπει να γίνουν και κάποιες πολιτικές επιλογές, οι οποίες θα γίνουν στο μέλλον από τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια τον συνομοθέτη. Όλα λοιπόν είναι στο τραπέζι, αλλά πιστεύω παράλληλα πως θα πρέπει να εξετάσουμε τις αναλλακτικέ λύσεις, οι οποίες, ε, τις οποίες περιέγραψε προηγουμένως κατά τα εισαγωγικά μου σχόλια και πιο συγκεκριμένα αυτές οι οποίες είναι πραγματική η υποκατάσταση της ε, κεροσύνης, γιατί, κυροζήνης με συγχωρείτε, ε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χαράξει την πορεία και είμαστε σοβαροί, είμαστε φιλόδοξοι και έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε τις ε, προϋποθέσεις έτσι ώστε να βρεθούν βιώσιμα υποκατάστατα καυσίμων για τον τομέα των, της και των αερομεταφορών. Εμείς θα πρέπει να καθοδηγήσουμε, εμείς θα πρέπει να χαράξουμε πορεία και πιστεύω πως χρειάζεται να έχουμε ε, μία δέσμη μέτρων με διάφορες εναλλακτικέ μέσω έρευνες, μέσω καινοτομία και το γεγονός πως κάθε αεροπλάνο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πετάει πολύ περισσότερα χιλιόμετρα από ό,τι χρειάζεται λόγω κατάτμισης του των εθέρων μας με αποτέλεσμα περισσότερες εκπομπές είναι απαράδεκτο και το γεγονός πως δεν έχουμε καταφέρει με πολιτική βούληση να ξεπεράσουμε την κατάτμιση και να πετύχουμε τους ενιαίους ευρωπαϊκούς ουρανούς ε, ας κάνουμε και μια προσπάθεια έτσι ώστε το αποτύπωμα του άνθρακα επιτέλους να εξεταστεί και να μειωθεί. Ο συντονιστής του ECR με ρώτησε θα συνεχίσει να αποτελεί μαζικό μέσο μεταφοράς του αεροπλάνου στο μέλλον. Ναι, σίγουρα. Γιατί μας εξασφαλίζει τη συνδεσιμότητα που είναι επίσης πολύ σημαντική. Κάποιος έρχεται από χώρες ε, εγώ, ε, εγώ προέρχομαι από χώρα που 30 χρόνια δεν είχαμε αυτή τη συνδεσιμότητα. Ξέρω πώς είναι. Αλλά για να συνεχίσουν οι μεταφορές να παίζουν αυτό το ρόλο πρέπει να έχει χώρο να αναπτυχθεί αλλά να μειώσει σημαντικά και το περιβαντολογικό του αποτύπωμα ο κλάδος. Οπότε ναι, θα συνεχίσουμε, αλλά για να έχουμε αυτό το περιθώριο θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά μέτρα που θα μας επιτρέψουν να δείξουμε πως είμαστε και εμείς συστρατευμένοι υπέρ της μείωσης των εκπομπών. Σίγουρα δεν απάντησα σε κάποιες ερωτήσεις. Να σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε, παρόλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που αντελήφθητε και σημειώσατε ότι υπάρχει σαφής πλειοψηφία εδώ στην ομάδα, στην Επιτροπή και τις πολιτικές ομάδες σε σχέση με την ρήτρα αποκλειστικότητας. Η Επιτροπή ελπίζω, αλλά και εμείς θα αναλάβουμε μια δράση συνολικά, συλλογικά σε σχέση με το Συμβούλιο, γιατί τελικά είναι και θέμα, είναι θέμα από τα κράτη-μέλη, όχι τις Επιτροπές. Και άρα σας διαβεβαιώ ότι εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στους διάφορους παράγοντες, ώστε να υλοποιηθεί αυτό το οποίο κατά πλειοψηφία αποφασίσαμε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δική μας η δυνατότητα να ρυθμίζουμε εσωτερικά τα ζητήματα αυτά. Περνώ στο επόμενο στάδιο της συζήτησης με τις ερωτήσεις στο σύστημα Catch the Eye, όποιος ενδιαφέρεται. Σημειώνω. Κύριε Βόλκεν, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία εδώ και για την ε, εισήγηση. Πρέπει να πω, πως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, πως είμαι απογοητευμένος από τις πρόοδους, η απουσία πρόοδων, που άλλωστε έχουν διεκδικήσει εκατοντάδες χιλιάδων νέοι, περισσότερη δηλαδή προστασία από την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη, μας το λένε συστηματικά. Μας λέτε ότι δεν είναι τέλειο το σύστημα. Πολύ σωστά, όχι μόνο δεν είναι τέλειο, είναι τελείως ατελές. Και έχουμε μια στρατηγική που μέσω του Κούρσια προσπαθεί να εισαγάγει, μάλλον να εισαγάγει την άρση συστημάτων που λειτουργούν σε επίπεδο περιφερειακό αρκετά καλά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρώ να δεχθεί. Μιλήσατε για την αποκλειστικότητα και αυτό με προβληματίζει κάτι. Αυτός ο κανόνα αυτός ο κανόνας λοιπόν αποκλειστικότητα σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει τη δυνατότητα να επιβάλλει φόρους κυροζήνης και αν ναι, θα ισχύει αυτό μόνο για τις εσωτερικές πτήσεις, μόνο για τις πτήσεις μεταξύ κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις πτήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτα κράτη και Τούμπαλεν. Ξέρω ότι εκεί είναι οι δυσκολίες στην υπόθεση αυτή. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ για την πολύ συγκεκριμένη αυτή ερώτηση και χωρί να θέλω βέβαια να σα ε, εκθέσω σε υπερβολικές πιέσεις, ζητώ από του συναδέλφου να μην διστάσουν να διατυπώσουν ακριβώ συγκεκριμένε ερωτήσεις. Ε, η κυρία Μπάουλης από του πράσινου, και υπενθυμίζω πως στη διαδικασία Καριστιάη ο καθένας έχει από ένα λεπτό για να διατυπώσει ερωτήσεις του. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον ομιλητή που μας περιέγραψε αυτή την κάκιστη συνθήκη της Κόρσιο που μιλάει για αντισταθμίσεις ε, ενώ χρειάζεται να έχουμε μηδενικές εκπομπές. Δεν είναι λύση δηλαδή για το μέλλον η Κόρσια. και μάλιστα δεν λύνει και προβλήματα σχετικά με, τους, ε, με τις εκπομπές στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας και τους υδρατμούς. Ούτε αυτή ούτε άλλες συμφωνίες. Ερωτώ λοιπόν, εάν ε, έχουν μελετηθεί σε όρους ε, αρρώσιμης γης ε, και άλλους οι εναλλακτικές λύσεις, Φερρυπίν βιοκαύσιμα που προτείνονται σαν αλλακτικά της κυροζήνης, γιατί αυτά θα έχουν συνέπειες. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εισαχθεί ένας φόρος κυροζήνης. Με το EBI ξέρετε ότι έχουμε αρχίσει να συλλέγουμε ε, υπογραφές γι' αυτό, για όλες τις ε, πτήση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο σύστημα ETS, όχι μόνο για να είναι πιο ακριβή η κυροζήνη και άρα οι αεροπορικέ μεταφορέ, αλλά και για να δώσουμε το καλό παράδειγμα στον υπόλοιπο κόσμο. Η κυρία Ντελή, SND. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω από το δεδομένο ότι έχουμε υπογραμμίσει πάντα πως, πως υπογραμμίζουμε πάντα πως όλοι οι τομείς, ε, όλοι οι κλάδοι πρέπει να συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών. Γιατί εδώ βλέπουμε πως κάποιοι τομείς φαίνεται να μην είναι διατεθειμένοι να, να μην εκτίθενται στην υποχρέωση να προσαρμόσουν τις εκπομπές τους. Εδώ λοιπόν που μας λέτε ότι το κόρσια είναι το μόνο μέσο που βασίζεται στην αγορά για τον περιορισμό των εκπομπών, αναιρείται ότι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρήση μέσων εργαλείων αγοράς αλλά και για τις εκπομπές. Και το ότι υπάρχει το Κόρσια δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει τίποτε άλλο ή ότι δεν κάνουμε κάτι άλλο. Και πάνω απ' όλα δεν σημαίνει ότι έχει λύσει τα προβλήματα και έχει επιτύχει τους στόχους που έχουμε ορίσει εμείς με το σύστημα ETS για την αεροπορία. Ένα-δύο ζητήματα επίσης που θα ήθελα να δώσει απαντήσεις ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι θα μπορέσει, θα επιδιώξει να κάνει μια ε, μέτριοπαθή απόπειρα για περιορισμό των εκπομπών η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Κόρσια, αλλά λίγα μόνο μπορεί να επιτύχει. Ωστόσο και πέραν της ε, εξουδετέρωσης εκπομπών, εγώ θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια και για τις διπλές καταγραφές. Αυτό πρέπει να το δούμε σε ένα παγκόσμιο σενάριο, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που μέτρο παρουσιάζεται ως λύση εκεί που τελικά δεν επιτυγχάνει τους στόχους για τους οποίους υποτίθεται πως έχει θεσπιστεί. Κυρία Λενουά Χρυνιού. Στα αγγλικά και στα γαλλικά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά. Είναι μεγάλη πρόκληση για την υγεία των Ευρωπαίων και των παιδιών τους. Ο περιορισμό των παγκοσμίων εκπομπών αντιλαμβανόμαστε ότι είστε επιφυλακτικός και ότι έχετε και υποχρέωση ενώ να μην, να μην ε, ε, ε, παραβιάσετε την αρχή της εμπιστευτικότητα σε σχέση με τι διαπραγματεύσει, Ωστόσο, είναι κρίσιμη σημασία και για λόγους διαφάνειας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων στην ΙΚΑΟ και σε σύντομους χρόνους να έρχεται ενώπιον του Κοινοβουλίου και να ενημερώνει για τις διαπραγματεύσεις αυτών, για τα αποτελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων. Σα Σας ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις? Όχι. Για την ανταλλαγή ενημέρωσης και εγγράφων. Βεβαίω όλε οι ομάδε υποστηρίζουν οποιοδήποτε μέτρο μπορείτε να εισαγάγετε για την ενίσχυση τη διαφάνεια. και την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ της υπηρεσίας σας και της Επιτροπής μας. Ευπρόσδεκτα όλα αυτά, γιατί κάθε ε, προσπάθεια για περισσότερη διαφάνεια θα μας ε, εξασφαλίσει και περισσότερη ε, αντίληψη, κατανόηση των όσων συμβαίνουν. Οπωσδήποτε θα είναι κάτι το καλό λοιπόν, μην διστάσετε. Απάντηση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις πρόσθετες ερωτήσεις. Στην, στο θέμα των εγγράφων, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι τα έγγραφα εργασίας είναι δημόσια και μπορεί κανείς να τα δει στο ιστοσελίδα της ΙΚΑΟ. Και άλλωστε θα τα βάλουμε και εμείς στο ενημερωτικό σημείωμα που θα σας ε, υποβληθεί το ταχύτερο, εφόσον εγκριθεί σήμερα από την Επιτροπή στη Συλλογική της Μορφή, όπως ελπίζουμε. Τώρα, μιλήσατε ξεκάθαρα για το θέμα της ε, αποκλειστικότητας, στο οποίο είχα δώσει νωρίτερα απαντήσεις, στο βαθμό που μπορώ. Στο στάδιο αυτό και για άλλη μια φορά σας ε, παρακαλώ να δείξετε κατανόηση ε, για το ότι είμαι, υποχρεω... δεσμεύομαι από τους κανόνες που διέπουν το έργο μου και ως εκ τούτου δεν μπορώ να δώσω περισσότερες απαντήσεις. Στο θέμα των φόρων και της αποκλειστικότητας, φορολόγησης και της αποκλειστικότητας. Η αποκλειστικότητα αυτή καθε αυτή δεν είναι ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με την ικανότητα επιβολής ενός φόρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτή είναι η πολιτική βούληση που θα εκφραστεί, θα είμαστε σε θέση να το πράξουμε χωρίς ε, κάποιο τύπου διακριτική μεταχείριση. Μετά, στο θέμα ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς μηδενικές εκπομπές, επίσης πιστεύω ότι επικρατεί συναντήληψη γενικά. Ωστόσο, τα μέτρα που ισχύουν σήμερα δεν αποδεικνύονται ικανοποιητικά και άρα φαντάζομαι θα συμφωνήσετε πως θα χρειαστούν τα μέτρα. Και πάλι εδώ τα βιώσιμα, όπως λέμε, καύσιμα για την αεροπορία θα έχουν κρίσιμο ρόλο για την ενίσχυση της ε, ε, πορείας προς τις μηδενικές εκπομπές. Χωρίς αυτά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε στις μηδενικές εκπομπές. Για το θέμα της διπλής προσμέτρησης ή καταγραφής, θα χρειαστούμε την ε, υποστήριξη και των διαπραγματευτών των Παρισιών, γιατί έχουμε το άρθρο 6 στη Συμφωνία των Παρισιών, με, την οποία, με το οποίο μπορούμε να καλέσουμε και την ΙΚΑΟ να αναλάβει τα σχετικά μέτρα. Η εξουδετερώση προβλέπεται σε κάθε συμφωνία, όχι μόνο στο Παρίσι, και πιο αυστηροί κανόνες ε, στο Παρίσι σημαίνουν και πιο αυστηρούς κανόνες για την Κόρσια. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να προχωρήσουν χέρι με χέρι εφόσον αυτή είναι η επιλογή μας. Νομίζω μέχρι εκεί θα, σταμα, θα πάω. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, de la part des, des coordinateurs, puisque nous avons encore... Οι συντονιστές έχουν κάποια άλλη ερώτηση ενδεχομένως. Θέλετε να επανέλθετε, Πέτερ Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χόλολάι διευκρινιστικά παρέθεσε τα λόγια της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και εμεί ε, τα ερμηνεύουμε. Αν θέλουμε να είμαστε ουδέτεροι ω προς το κλίμα μέχρι το 2050 και ε, από την άλλη να τονίσουμε τη σημασία του Κόρσια ως σημαντικό εργαλείο, Πρέπει να πω ότι το Κόρσια δεν μειώνει καθόλου τις εκπομπές στις αερομεταφορές. Απλά αντιστάθμιση γίνεται με πολύ θολά μέτρα και έτσι θα έχουμε αύξηση και μάλιστα ραγδαία αύξηση των ε, εκπομπών. Εάν θέλουμε να είμαστε ουδέτεροι ως προς το κλίμα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα στον τομέα του ατσαλιού, στον τομέα άλλων βιομηχανιών θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον Γενικό Διευθυντή. Δεν θα πρέπει να πούμε με πολύ πιο ξεκάθαρα λόγια ότι το Κόρσια είναι κακό. Είναι δηλαδή πολιτικά απαραίτητα... μάλλον καταλαβαίνω ότι είναι πολιτικά απαραίτητο να συνεχίσουμε τις εργασίες μας στην ΙΚΑΟ, αλλά δεν θα πρέπει να πούμε με πολύ πιο καθαρά λόγια ότι είναι κακό το Κόρσια. Ωραία, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από το S&D. Όχι. Από το Renew. Όχι. Πράσινη. Ναι, θέλω να πιέσω λίγο τον κύριο Χολουλάη όσον αφορά τη νομική πτυχή που έθιξε ο συνάδελφος ο κύριος Βίλκεν, διότι δεν μπορεί να κρύβεται κανείς πάντα πίσω από ε, τους κανόνες ε, Υπάρχει πάντα μια νομική ανάλυση. Δηλαδή, αν υιοθετηθεί αυτό, τι θα σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Εάν έχουμε ένα σύστημα εμπορία εκπομπών για τις εσωτερικέ πτήσει και η ΚΑΟ πει ότι μια πτήση ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία είναι ε, διεθνή πτήση και εμεί πούμε ότι όχι είναι εσωτερική. Αυτό νομικά πώ ε, ερμηνεύεται. Και επίσης μπορούμε να σταματήσουμε το ρολόι, να πούμε δηλαδή ότι αν δεν αρκούν όλα αυτά θέλουμε να αναλάβουμε δράση όσον αφορά τις πτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτες χώρες και αντιστρόφως. Αυτό θα είναι δυνατό όταν θα έχει υιοθετηθεί αυτή η πρόταση. Αυτό ε, έχει να κάνει με νομική ανάλυση. Δεν έχει να κάνει με την ε, υποχρέωση εμπιστευτικότητας που έχετε στο πλαίσιο του ΙΚΑΟ. Ε, θέλουμε αυτή την απάντηση, Αλλιώ δεν μπορούμε εμεί να διαμορφώσουμε θέση. Και μην κρύβεστε πίσω από την ΙΚΑΟ. Άλλε ομάδε uh, Άλλες ομάδες θέλουν να πάρουν το λόγο. ID. Είστε μέλος του ID, όχι. Ε, στους συντονιστές δίνω το λόγο μόνο. ECR. Γκουε. Όχι, δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Ωραία. Δύο τελευταίες παρατηρήσεις λοιπόν που ακούσαμε από το ΕΛΚ και τους πράσινους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και πάλι για τις δύο αυτές δύσκολες ερωτήσεις. Ουδετερότητα μέχρι το 2050. Ε, Νομίζω ότι είναι σαφέ ότι αυξάνεται το επίπεδο φιλοδοξίας και σε αυτό αναφερόμουν και άλλωστε είναι πολύ ε, καθαρό το μήνυμα της ε, ε, εκλεγής σας Προέδρου. Όσον αφορά το Κόρσια, δεν θα πω ότι είναι κακό. Θα πω ότι είναι ατελές. Συμφωνήθηκε το 2016 και απομένει να το εφαρμόσουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Όταν όμω σκεφτόμαστε την Ευρώπη, ποτέ δεν θεωρήσαμε το Κόρσια να είναι το μόνο εργαλείο μα διότι κάνουμε πολλά άλλα πράγματα. Πάντα μιλούσαμε για μια δέσμη μέτρων και το Κόρσια ήταν ένα στοιχείο σε αυτή τη δέσμη. Είναι σαφές ότι αν θέλουμε να κινηθούμε με την φιλοδοξία που έχουμε εκφράσει, τότε είναι σαφές ότι θα πρέπει να κινηθούμε με διάφορα μέσα. Ταυτόχρονα το με το Κόρσια θα έχουμε ουδέτερη ως προς τις εκπομπές ε, ανάπτυξη. Εάν όμως δεν έχουμε το Κόρσια, αν δεν έχουμε κανένα παγκόσμιο πρόγραμμα, τότε ναι, μπορούμε να κάνουμε τέλεια δουλειά στην Ευρώπη, αλλά σε έναν ε, πολύ... Ε, σε έναν καθόλου τέλειο κόσμο. Είναι απαραίτητο ένα παγκόσμιο σχέδιο, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουμε μια παγκόσμια πρόκληση. Γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε με το Κόρσια ώστε να γνωρίζουμε ότι οι βασικές ε, χώρες ε, που αναπτύσσονται τώρα να δεσμεύονται από τους κανόνες του Κόρσια και θα είναι δύσκολος ο δρόμος μπροστά μας, ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Φυσικά, το κόρσια και το σύστημα εμπορίας εκπομπών, όπως είπα και νωρίτερα, θα αναθεωρηθούν. Στο μέλλον ε, και η ανάλυση συνύπαρξη στην οποία αναφερθήκατε και εσεί, κύριε Πρόεδρε, είναι μια δουλειά που συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω ότι θα είναι αδύνατον να συνυπάρχουν τα δύο αυτά προγράμματα. Ε, τούτη τη στιγμή όμως δεν μπορώ να σας παρουσιάσω στοιχεία συγκεκριμένες ανάλυσης, διότι δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου και δεν θα ήθελα να ε, να παρατεθούν λάθος τα λόγια μου αργότερα. Αλλά πάντως, ε, εν καιρό, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, θα σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε έτσι την πρώτη σημερινή ακρόαση. Προτείνω πέντε λεπτά διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά. Colleagues, oh wow, that's loud. Okay, uh, thank you very much. Um, colleagues, the uh, our chair has uh, vacated to. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο συνάδελφος, ο πρόεδρος ε, έφυγε γιατί έχει μια άλλη συνεδρίαση. Αναλαμβάνω εγώ λοιπόν. Και θα σας παρακαλέσω λίγο πιο ήσυχα. Έχουμε λοιπόν τώρα ανταλλαγή πληροφοριών ε, για τα θέματα που θα αφορούσαν το REACH γενικότερα ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Της δίνω 10 λεπτά. Πέντε λεπτά έκαστος, μια και είστε δύο. Κύριε Σπιτινέλη, Grow. Και μετά Σεντάουσκας, Envy. Κύριε Πετινέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να ασχολείται με τα χημικά πριν 50 χρόνια και Έχουμε επιδείξει αφοσίωση απέναντι στην προστασία της ε, ανθρώπινης υγείας ε, και του περιβάλλοντος, καθώς και της ομαλής λειτουργίας ε, της εσωτερικής αγοράς. Το παρόν θετικό πλαίσιο καλύπτει τα χημικά, τη, τη θέση του καταναλωτή, τα λιπάσματα, τα απόβλητα και τα ύδατα. Από τη στιγμή που παράγονται τα χημικά, τη χρήση τους και την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον. Και ο έλεγχος καταλότητας απαντάει σε τρία βασικά ερωτήματα. Τι έχει πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των χημικών. Πάνω από 40 οδηγίες ε, και κανονισμοί που περιέχουν ε, μία ή περισσότερες διατάξεις ε, για τα χημικά, πώς λειτουργούν σε συνδυασμό η μία με την άλλη και ποια είναι τα ισχυρά σημεία και οι αδυναμίες της νομοθεσίας για τα χημικά και ο έλεγχός μας εξετάζει όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξετάσαμε επίσης ε, την εφαρμογή και επιβολή των κανόνων από τα κράτη-μέλη ο έλεγχος καταλληλότητας ε, συμπληρώνει ε, την αξιολόγηση της ε, νομοθεσίας REACH που δημοσιεύτηκε πέρσι. Και αυτές οι δύο αξιολογήσεις καλύπτουν το σύνολο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χημικά. Ο έλεγχος καταλληλότητας καταλήγει ότι είναι κατάλληλη η νομοθεσία για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τα χημικά. Κατοπτρίζει 50 χρόνια συνεχών προσπαθειών και η προστιθέμενη εξέλιξη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο στον τομέα των χημικών είναι σαφώς υψηλή. Και η πολιτική μας και η διαδικασία λήψη αποφάσεων αποτελεί ε, έμπνευση για πολλές άρες χώρες. Η λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εναρμόνιση και τα κοινά πρότυπα ε, εξασφαλίζουν ίσα επίπεδα προστασίας ανθρώπων και του περιβάλλοντος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έτσι ενισχύεται η εσωτερική αγορά και έχουμε ανταλλαγή γνώσεων και πόρων. Όμως, εντοπίσαμε πεδίο, ε, περιθώριο βελτίωσης ε, κατά την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας καθώς και την ικανότητά μας για συνεργασία. Όσον αφορά ε, αντικείμενα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ε, δημόσιες αρχές θέλουν να εξασφαλίσουν προστασία του καταναλωτή, αλλά και δίκαιο ανταγωνισμό ανάμεσα σε εταιρείε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τρίτες χώρες. Αυξάνεται συνεχώς ο όγκος των προϊόντων που πολλούνται ε, στο διαδίκτυο και οι οικονομικοί φορείς ε, δεν, ε, δεν μπορούν πάντα να ε, εγγυηθούν ότι τα προϊόντα που πολλούνται στις πλατφόρμες τους δεν περιέχουν επικίνδυνα χημικά. Επίσης, συχνά είναι ελλειπής η αξιολόγηση κινδύνου των προϊόντων αυτών οι οικονομικοί φορείς πρέπει να κατανοούν τους κανόνες και να παρακολουθούν τις αλλαγές στην νομοθεσία. Σαφήνεια των κανόνων διευκολύνει και αυξάνει την συμμόρφωση με τους κανόνες. Οι οικονομικοί φορείς συχνά δυσκολεύονται περισσότερο ε, στο θέμα αυτό λόγω διαφόρων περιορισμών. Υπάρχουν κάποιες ε, ε, ατέλειες ε, στις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται από επιστημονικούς φορείς. Ε, οι κίνδυνοι αυτοί προκύπτουν από την ομαδική αξιολόγηση χημικών αντί να γίνεται ξεχωριστή αξιολόγηση για κάθε είδος. Επίσης, εξετάζουμε την παραγωγή χημικών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία πρόκληση αποτελεί η αυξανόμενη ψηφιοποίηση και ο αυξανόμενος εστιασμός στην βιωσιμότητα. Έτσι μπορεί να αμφισβητηθεί η κορυφαία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν στο μέλλον για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση μπορούμε να βασιστούμε στην ανεπτυγμένη βιομηχανία χημικών, στην εσωτερική αγορά που είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο που προτείνει τους καταναλωτές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους επιτρέπει να ε, λαμβάνουν περιστατωμένες αποφάσεις. Οι καταναλωτές ε, έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα προϊόντα που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα εισαγόμενα και μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερη χρήση των ευφυών τεχνολογιών. Ε, έτσι θα μπορούν οι καταναλωτές να λαμβάνουν καλές αποφάσεις. Ε, μπορεί να βελτιωθεί ο τρόπος που μεταφέρουμε πληροφορίες στους καταναλωτές και σε οικονομικούς φορείς σε όλη την αλυσίδια προμήθειας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου. Παρακαλώ. Thank you, In terms of protection of health and environment... Για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αυτό αποδεικνύει πως η σχετική νομοθεσία μας έδωσε πολλές επιτυχίες. Για παράδειγμα, η έκθεση των πολιτών ε, στα βαρέα μέταλλα, για παράδειγμα, βενζινοειδή, ε, και άλλες χημικές ενώσεις που έχουν μειωθεί σημαντικά. Παρ' όλα αυτά είναι πολλές ε, ανησυχητικές ε, παράλληλες εξελίξεις με προβλήματα γονιμότητας για τους ε, άνδρες στην ε, Ευρώπη, ε, νευρολογικές ασθένειες, κάποια είδη καρκίνων. Όλα αυτά έχουν πολύπλοκους και πολλαπλούς παράγοντες που τα επηρεάζουν ε, και η δική μας αξιολόγηση μας οδηγεί στο εξής. Οι προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι πρώτον τα νομοθετικά μέτρα να είναι συνεκτικά μεταξύ τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη προστασία και κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες. Όσο δεν υπάρχει οριζόντια προσέγγιση, μπορεί οι ευάλωτες ομάδες να μην προστατεύονται με ισότιμο τρόπο. Ε, για παράδειγμα, σε κάποιες κατηγορίες ε, όπου οι ανώτατες τιμές δεν συμπίπτουν. Επίσης, αναδυόμενοι κίνδυνοι. Και εδώ χρειαζόμαστε ιδιαίτερη προσοχή. Και ίσως εδώ θα έπρεπε να έχουμε ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης στην Ευρώπη. Τρίτον, οι τρέχουσες γνώσεις που έχουμε για την έκθεση στις βλαβερές χημικές ουσίες και ο αντίκτυπος αυτής της έκθεσης για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον δεν είναι αρκετές. Χρειαζόμαστε περισσότερα. Πρέπει να παρακολουθούμε τις ε, βλαβερές ουσίες και στα πλαίσια της οικονομίας του διαμοιρασμού. Πέμπτον, δεν έχουμε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχουμε προχωρήσει σε υποκατάσταση των βλαβερών χημικών ουσιών ε, μέσω της τρέχουσας νομοθεσίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πιο στενά τι γίνεται με τα νέα χημικά που μπαίνουν στην οικονομία μας το μέλλον, όπως είπε και ο κύριος Πετινέλη. Ίσως η νομοθεσία μας εδώ να είναι η πιο φιλόδοξη στον κόσμο και είναι α, πραγματικά υψηλή η προστασία που προσφέρουμε στους πολίτες μας και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Όμως υπάρχουν πάρα, πολλά, πάρα πολλές προσ προκλήσεις. Τον Ιούνιο έγινε μια υψηλό επίπεδου ε, συνεδρίαση ε, για τον έλεγχο καταλληλότητας ε, για τα εντός ρίτς τα περασμένα χρόνια, όπως επίσης και για μια νέα αξιολόγηση. Όλα αυτά θα τροφοδοτήσουν τη συζήτηση για τη συζήτηση στο μέλλον νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το έχει συμπεριλάβει, όπως επίσης και το θέμα με τους διαταράκτες, αλλά και με τη μηδενική ρήπανση. Άρα λοιπόν η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη βάση για να σχεδιάσει και το μέλλον της, αλλά και τα μέτρα για την πολιτική για τα χημικά στην Ευρώπη. Okay, thank you very much. Uh, we have... Σας ευχαριστώ. Τρεις συναδελφές του το λόγο μέχρι τώρα. Για πείτε μου. Πέτερ Λίζα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι σημαντικό βέβαια το ριτς για να προστατεύσουμε τους πολίτες από τα επικίνδυνα χημικά. Και επίση είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσει για τέτοια θέματα, ώστε να μην γίνονται, να μην ρυθμίζονται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Ξέρουμε ότι η βιομηχανία χημικών προϊόντων δεν έδειξε μεγάλη χαρά στην εισαγωγή του Ριτς. Τώρα όμως μας λένε πως να, με το Brexit το σημαντικότερο από όλο το Ριτς εξακολουθεί να ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο και άρα δεν θα έχουμε διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής ή ε, παντιοτρόπως ε, προβλήματα γραφειοκρατικού χαρακτήρα να ξεπεράσουμε ε, με την εισαγωγή του Brexit στον τομέα των χημικών. Είναι σημαντικά όλα αυτά λοιπόν. Μας λέει η Επιτροπή ότι δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με απολύτο τρόπο. Ε, αν μια ουσία βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται σε μια διαδικασία παραγωγής, μπορούμε να ξέρουμε ότι είτε δεν προξενεί, δεν απειλεί την υγεία του ανθρώπου, είτε απαγορεύεται. Και αυτό μπορούμε να το δείξουμε με κάποια παραδείγματα που νομίζω μπορούν να, να, να είναι χρήσιμα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το χρώμιο καταρχάς, που μάλιστα με μια αμφιταλαντευόμενη πλειοψηφία μπορέσαμε να περάσουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγορεύοντα, απαγορεύοντας όπως θέλανε πολλοί, το οποίο όμως δεν έχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία παρά μόνο ε, ανάλογα με τον τρόπο στον οποίο χρησιμοποιείται σε μια διαδικασία παραγωγής η οποία θα μπορούσε ε, να ξεπεραστεί από τους παραγωγούς, ε, εφόσον απαγορευόταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εισαγωγές από τρίτα κράτη που δεν θα είχαν εξίσου αυστηρές προδιαγραφές. Στα μικροπλαστικά επίσης. Λέμε ότι χρησιμοποιούνται τα μικροπλαστικά και αυτά πρέπει να απαγορευθούν οπουδήποτε και αν χρησιμοποιούνται. Αυτό θα έχει όμως ε, πολύ ριζικές συνέπειες. Όπως σε παραδείγματι στο τεχνητό γκαζόν που χρησιμοποιείται σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Η εναλλακτική που θα είχαμε αν απαγορευόταν αυτό θα ήταν και επικίνδυνη για την υγεία των αθλητών και άρα δεν θα μπορούσαν να ασκήσουν το άθλημά τους. Πρέπει επομένως να αναζητούμε εναλλακτικέ να επιτρέπουμε μακρές περιόδους προσαρμογή ώστε να μπαίνει και η τεχνολογία στη διαδικασία αυτή προσαρμογής για να δώσει νέε λύσεις και γι' αυτό καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην έχει τόσο απόλυτη συμπεριφορά και αυστηρή όταν ε, θεωρεί ότι υπάρχει λόγος να ε, περιοριστεί η χρήση μια ε, ουσίας από την οποία ενδέχεται να προκύπτει κίνδυνος από την έκθεση για τον άνθρωπο, αλλά να αφήνει ένα περιθώριο για προσαρμογή. Ευχαριστώ κυρία Χάζενκαμπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας διαφώτισε. Έχουμε εδώ λοιπόν να κάνουμε με ένα κείμενο ε, ομπρέλα ε, το οποίο θα πρέπει να απαγορεύεται ε, μεν να απαγορεύει μια ουσία, να παραδείγματι αντιληφθούμε ότι μια ουσία επικίνδυνη μπορεί να μπει μέσα στο γάλα που πάει στο μπιμπερό, ή στο μπιμπερό το ίδιο των παιδιών σαν ε, χημική ένωση, να απαγορεύεται και ταυτόχρονα να ελέγχεται ώστε να μην μπαίνει πουθενά αλλού σε μια τροφική αλυσίδα ή γενικά να καλύπτεται από όλα τα νομοθετικά κείμενα. Αυτό ισχύει και για τα ζώα φυσικά και γι' αυτό οι ενώσεις προστασία των ζώων προσπαθούν να επιβάλλουν μια απαγόρευση για, για τις ε, κλινικές δοκιμές εις βάρος ζώων. Η ανάλυση όμως θα πρέπει να αφορά τον κίνδυνο και για τον παραγωγό, ώστε και αυτός να αναλάβει τις ευθύνες των επιλογών του και να ε, καταστεί ταυτόχρονα η οικονομική μας δραστηριότητα και οι επιλογές μας οικονομικές πιο διαφανείς. Πρέπει επικίνδυνες ουσίες να απαγορευθούν Πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει ο κλάδος, το είπε και ο καθηγητής Ρουτλάν στην, ε, ε, στο σεμινάριο που κάναμε για τις χημικές ε, ουσίες, για τις επικίνδυνες ουσίες. Μας είπε λοιπόν ότι ακόμα δεν υπάρχουν ουσιαστικέ προτάσεις και πρέπει αυτό να αλλάξει. Ευχαριστώ κύριο Σαντεχούζα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που εθέσατε και το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Είναι πολύ σημαντικό για μας να συζητήσουμε την ε, χημική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ακούσαμε και πριν, πιστεύω και εγώ ότι υπάρχει ανάγκη για πιο αυστηρή και καλύτερη νομοθεσία για τα χημικά και στον τομέα του Ρίτσα, παρότι δεν συζητάμε αυτό αυτή τη στιγμή. Διότι αν δεν είμαστε αρκετά γρήγοροι στις αντιδράσεις μας όσον αφορά μονομένες ουσίες, όταν ε, συμβαίνει κάτι, θα δούμε ότι τα κράτη-μέλη θα ε, λαμβάνουν μεμονωμένες αποφάσεις ε, και το καταλαβαίνω αυτό. Για παράδειγμα, η νέα δανέζικη κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει τις κάποιες ουσίες στο χαρτί ψησίματος που περνάνε στα τρόφιμα και που βλάπτουν μεταξύ άλλων ε, τα έμβρια. Και αν δεν το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκαίρως ε, τα κράτη-μέλη θα λαμβάνουν αποφάσεις ε, όταν βλέπουμε νέες μελέτες για μεμονωμένες ουσίες που να βλάπτουν την υγεία. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να αντιδράμε όχι σε 5 ή 10 χρόνια, αλλά τώρα. Και αν δεν καταφέρουμε να χειριστούμε το θέμα αυτό καλύτερα, θα έχουμε μεμονωμένε απαγορεύσει στα κράτη-μέλη και θα καταστρέψουμε την εσωτερική αγορά. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για καλύτερο χειρισμό. Συμφωνώ ότι έχουμε την καλύτερη χημική νομοθεσία στον κόσμο και ότι προστατεύουμε καλύτερου καταναλωτέ ε, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο, αλλά ε, υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που εξετάζετε το θέμα αυτό και χαίρομαι που ε, η νέα πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε το θέμα αυτό στο πρόγραμμα εργασία τη. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολιτική χημικών που να μα επιτρέπει πιο γρήγορη αντίδραση όταν διαπιστώσουμε ότι κάποιε μεμονωμένε ουσίες μπορεί να έχουν κάποιο κίνδυνο όταν έρχονται σε επαφή με αυτέ οι πολίτε μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρίς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε όντως ε, την πιο φιλόδοξη στα θέματα των χημικών ουσιών ε, νομοθεσία στον κόσμο. Επισημάνθηκε αυτό ήδη. Και μπορούμε να είμαστε νομίζω όλοι με το δίκαιο μας υπερήφανοι γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποια σημεία τριβής με την προηγούμενη επιτροπή έγινε λόγο σε παραδείγματα για του ενδοκρινικού διαταράκτε και με ικανοποίηση ακούω ότι ε, από τον εκπρόσωπο τη επιτροπή ότι είναι εξελίξη ένα απολογισμό ε, συνεπειών. Το θέμα της γλυφοζάτης, η ενίσχυση της νομοθεσίας που ζητούμε για τα ζυζονιοκτώνα ε, είναι εν εξελίξη, είναι σε εκκρεμότητα. Ε, περιμένω καλές εξελίξεις και σε αυτό. Ο κύριος Κουτσί και τον εκπροσωπώ σήμερα γιατί δεν μπόρεσε να έρθει και στη συγγνώμη. Μου ζητεί να σας μεταφέρω τις ερωτήσεις του και στα αγγλικά μάλιστα. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι υπάρχουν μελέτες για πλαστικά σε διάφορα αισθήματα, πλαστικά που φτάνουν μέχρι και στα τρόφιμα μας και μπορεί να είναι ε, καρκινογόνα, να έχουν διαταρακτική των ορμονών λειτουργία ή να γεννούν άλλα προβλήματα. Πότε θα υπάρξει μια μελέτη και πότε θα δούμε μια φιλόδοξη και γενική ε, νομοθεσία η οποία θα δώσει αποτελεσματική λύση. Ο συνάδελφος λοιπόν μου μας λέει ότι ενημερώθηκε πως μια τέτοια έρευνα μελέτη θα δημοσιευθεί το 2020 και ζητεί επιβεβαίωση. Επίσης υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία ε, έχουν παρεμποδίσει την ε, επίτευξη αποτελεσματικών στόχων ε, για τα θέματα αυτά και μπορεί να τα εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα παιχνίδια ή για ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς αντιμετωπίζει την απουσία υλοποίηση από, από αυτά τα κράτη-μέλη. Και επίσης, παρότι είναι η νομοθεσία μας εύρωστη, δεν βλέπουμε μία τάση μετάβασης προς πιο αθώα ή λιγότερα επικίνδυνα ε, χημικά. Και έτσι έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά, 60 και 40% αντίστοιχα για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία χημικών που χρησιμοποιούνται και που είναι ε, υπεύθυνα για χιλιάδες προεμούς θανάτους και για απώλεια βιοπικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει κάνει για να αντιμετωπίσει, να ανατρέψει αυτήν την τάση. Ευχαριστώ. Συνήθως έχουμε ένα μακρύ κατάλογο ερωτήσεων και μετά δίνουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή ο κατάλογος είναι αρκετά σύντομος αυτό το γύρο και έχω ακόμα κάποια ονόματα, τρεις συνάδελφοι θέλουν κάτι να ρωτήσουν και επειδή είναι πολύ λεπτομερεί οι ερωτήσεις, θέλω να εξασφαλίσω πως οι απαντήσεις θα δοθούν. Έχουμε χρόνο Μετά τους επόμενους τρεις λοιπόν θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά εκ νέου σχόλια. Παρακαλώ πολύ. Η κυρία Πάουλους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την δουλειά που κάνετε σε αυτή τη διαδικασία refit και δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει, αλλά για όσους κοίταξαν το έγγραφο ε, έχετε εξετάσει πολύ βαθιά. Είχατε τέσσερα χρόνια, αλλά εμείς θέλουμε και παραπάνω στοιχεία και για τους ε, ενδοκρινολογικούς διαταράκτες και για τα τις βλαβερές χημικές ουσίες και για τη βιοπικολότητα. Είπατε πως υπάρχει η αρχή της πρόληψης, αλλά δεν εφαρμόζεται ολοκληρωτικά. Επίσης, ουσίες οι οποίες είναι ανισχυτικές σε, ε, σε καθημερινά προϊόντα, ε, προβλήματα για τον καταναλωτή, η οικονομία του, κυκλική οικονομία, με συγχωρείτε, ε, εντομοκτώνα τα οποία παραμένουν σε κυκλοφορία γιατί τα κράτη-μέλη δεν σέβονται τις ημερομηνίε. και σορευτικές συνέπειες, δράσεις για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, Εκπλήσουμε λοιπόν από τα συμπεράσματα ή από το σχέδιο δράσης, γιατί δεν βρήκα ποιο είναι το όραμά σας για μια βιώσιμη νομοθεσία για τα χημικά που να λαμβάνει υπόψη και την ανθρώπινη υγεία και τη διατήρηση των φυσικών πόρων που αποτελούν και τη βάση επιβίωσης ημών. Μοιάζουν όλα αυτά να είναι πιο ε, λιγότερο ενισχυτικά από την κοινή αγορά. Αυτό για μένα δεν είναι σωστό. Μιλήσατε για έλλειψη επιστημονικών γνώσεων. Ωραία, τι θα κάνετε λοιπόν, θα λάβετε δράση για μη τοξικό περιβάλλον. Έχετε περιγράψει κάποιο πλαίσιο και στρατηγική. Θα έπρεπε ήδη το 2018 να έχει καταστρώσει κάτι αντίστοιχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πότε λοιπόν. Τέλος. Στρατηγική για μηδενικούς ρήπους. Η κυρία Βαντερ το έχει υποσχεθεί. Σίγουρα έχετε κάποιο σχέδιο δράση. Πότε θα το παρουσιάσετε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νόβακ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας πω τι μου είπαν ε, οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα στη Γεωργία. Όλοι αναφέρουν πως ικανοποιούνται πλήρως από την νομοθεσία για τα φαρμακευτικά παρασκευάσματα έχουν εκπαιδευτεί, τους έχουν δώσει περαιτέρω ε, πληροφορίες και η χνηλασιμότητα έχει βελτιωθεί. Αυτά είναι τα θετικά πρόσημα, αλλά έχουμε και κάποιες αρνητικές ε, πτυχές, κυρίως την ε, διαχείριση των αποβλήτων όπως επίσης και στην αποθεματοποίηση των αποβλήτων. Εκεί δεν υπάρχει συστηματική καταλογοποίηση και είναι και διαφορετικοί οι δείκτες μέτρηση που χρησιμοποιούνται. Άλλες φορές είναι οι κιλά, άλλες υπολογισμό γίνεται σε κυβικά μέτρα, σε λίτρα, σε τόνους καμιά φορά, οπότε αυτό δεν έχει ε, ενοποιηθεί. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει προβλέψει κάποια νέα δράση για τη διαχείριση των αποβλήτων και για την ε, αποθήκευση των αποβλήτων. Και η κατηγοριοποίηση αυτών θα γίνει με πιο συστηματικό και ενοποιημένο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ με τη σειρά μου κάποια πράγματα. Οι συνάδελφοι ήταν πολύ ευγενικοί μαζί σας και εγώ θα παίξω τον κακό αστυνομικό. Γιατί εγώ απογοητεύτηκα. από τον έλεγχο καταλληλότητας το μόνο που καταλαβαίνει κανείς ότι όλα πάνε καλά. Η εντύπωση είναι πως εντάξει υπάρχουν προβλήματα, αλλά γενικότερα η νομοθεσία είναι καλή. Κατάλληλη λοιπόν, με υψηλό επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό που βλέπουμε είναι μια αύξηση των σοβαρών ασθενειών στην Ευρώπη και συνδέεται αυτή η αύξηση με τα χημικά. Εύκολα θα μου απαντήσετε. Αν όλα λειτουργούν τόσο καλά, πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί πως οι ασθένειες που συνδέονται με την έκθεση χημικά αυξάνονται στην Ευρώπη. Ενδοκρινολογικοί διαταράκτες, για παράδειγμα, και δημόσια υγεία. Και ρωτώ το εξή επίση, γιατί δεν έχει δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αυξήσει τα επίπεδα προστασία κατά των διαταρακτών, έτσι ώστε όλοι καλύπτονται. Να, τα πλαστικά, τα υφάσματα, το πόσιμο νερό, ξέρουμε πως δεν προστατεύεται αποτελεσματικά ο πολίτης. Κινδυνεύει η υγεία του και θέλουμε από σας πιο αποτελεσματική δράση. Και για τη συμμόρφωση. Μία πρόσφατη μελέτη του Γερμανικού Ινστιτούτου για την Αξιολόγηση Κινδύνου και το Περιβαλλοντικό Ινστιτούσο, το 1 τρίτο ε, των ε, χημικών που παρασκευάζονται ή εισάγονται στην Ευρώπη το 2010 καταπατούν το ευρωπαϊκό δίκαιο που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν από τη βλαβερή έκθεση το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Μόνο 31% ήταν νομικά σύμμορφα. Η νομοθεσία REACH υποχρεώνει τις εταιρείε να ε, αναφέρονται για το κατά πόσο οι ουσίες τους δημιουργούν ε, οποιοδήποτε ε, οποιοδήποτε προβλήματα στην ανθρώπινη γονιμότητα, στην, ε, στις ασθένειες παιδικές, στα νευρολογικά, στα ορμονικά, στην τοξικότητα. Γιατί λείπουν αυτές οι πληροφορίες. Τέλος. Οι σοσιαλιστές ρωτούν πότε θα παρουσιάσετε επιτέλους την στρατηγική που αναμένουμε τόσο καιρό για το μη τοξικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ένα καθαρό περιβάλλον. Είναι πολύ εύκολο να μιλά κανείς για το θέμα αυτό. Αλλά θέλουμε, εκτός από λόγια, δράσεις για να ενισχύσουμε το επίπεδο προστασίας του Ευρωπαίου πολίτη και του, Ευρωπαίου, και του Ευρωπαϊκού με συγχωρείτε περιβάλλοντος. Πολύ λεπτομερείς ερωτήσεις αλλά θα ήθελα να απαντηθούν. Δεν λέω πως δεν θα απαντήσετε, αλλά αυτό που γίνεται συχνά στις συναντήσεις αυτές είναι πως έχουμε μια τεράστια λίστα ερωτήσεων και πολύ λίγο χρόνο για να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφού λοιπόν έχουμε χρόνο, καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στα όσα ακούστηκαν μέχρι στιγμής και για τους επιπλέον ε, ομιλητές στον επόμενο γύρο θα δώσω προτεραιότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν μιλήσει. Παρακαλώ λοιπόν, αν μετά θεωρήσετε πως δεν απαντήθηκε η ερώτησή σας, σηκώστε το χέρι σας για να λάβετε συγκεκριμένη απάντηση. Κύριε Πετινέλη, κύριε Σαντάουσκας, 10 λεπτά ο καθένας, 10 λεπτά και οι δύο μαζί και μετά ερωτήσεις. Yes, thank you. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για σαν του κυρίου Λίσσα. Ακριβώς αυτή θα ήθελα να σας πω. Είναι η λειτουργία του κανονισμού REACH. Προσπαθεί να λάβει υπόψη όλες τις ε, πτυχές. Και γι' αυτό υπάρχει και η Επιτροπή Αξιολόγηση Κινδύνου, αλλά και η ΣΕΚ που αξιολογεί τον οικονομικό και κοινωνικό, τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Κατόπιν των εκθέσεων αυτών των δύο επιτροπών λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση όλες τις πληροφορίες που θα τις παράσχουν τις σχετικές αποφάσεις. Και έτσι προσπαθώντας βέβαια να δώσει την καλύτερη λύση με την ε, καλύτερη ισορροπία που βέβαια δεν είναι σαφές ε, πάντα τι σημαίνει για όλους γιατί μπορεί η καλύτερη ισορροπία να είναι διαφορετική για τον καθένα. Στα χρωμιώδη παραδείγματα ε, είδαμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί, διαφορετικές αρχές και κανόνες και για το Κοινοβούλιο. Στην υλοποίηση. Είναι μια πρόκληση η υλοποίηση ασφαλώς καθώς η νομοθεσία είναι περίπλοκη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που καλούνται να υλοποιήσουν, αλλά τον έλεγχο της επιβολής τον έχουν τα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν τι γίνεται, έχουμε κανόνες πιο απλούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό επιδιώκουμε να έχουμε, ώστε να είναι μικρότερη η επιβάρυνση όταν πρέπει κανείς να αξιολογήσει τους κινδύνους μιας ουσίας ή όταν πρέπει η αξιολόγηση να μεταγραφεί σε δεδομένα από τα κράτη. Ε, πολιτικό πρόγραμμα και θεματολόγιο της Επιτροπής, της Νέας Επιτροπής θα είναι, από ό,τι λέει η Πρόεδρος, ε, ένα πιο απλό σύστημα αλλά και πιο αυστηρή, αυστηρές κυρώσεις για όσους ε, παραβιάζουν ή υποβαθμίζουν τους ε, κανόνες η διαδικασία, ξέρετε, για την εγκαθίδρυση της Νέας Επιτροπής είναι σε εξέλιξη, άρα δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε πιστωρές λεπτομέρειες, γιατί δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί αυτές και όχι γιατί δεν θέλουμε να σας τις δώσουμε. Ε, είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η διαδικασία και η πρόεδρος έχει αναλάβει αυτές τις δεσμεύσεις για τα τρόφιμα και το υλικό αυτό, τα, τα, τις ουσίες αυτές, είναι σε εξέλιξη μία μελέτη που θα εξετάσει και ένα πιο ε, ουσιαστικό τρόπο αξιολόγησης με μια διαδικασία που ούτως ή άλλως ήδη είναι ε, πολύ απαιτητική και προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο ε, προστασίας. Φυσικά πάντα μπορεί να γίνει πιο απαιτητική, αλλά δεν ξεκινάμε και από το μηδέν. Και επίσης μια εξωτερική μελέτη θα ολοκληρωθεί σύντομα, μια μελέτη η οποία θα μας δώσει πιο λεπτομερή στοιχεία και θα δημοσιευθεί σύντομα. για τα μέσα. Βεβαίως αυτά σχετίζονται και με την διαθεσιμότητα των πόρων. Ε, οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών πρέπει να προχωρεί με βάση την ε, δειγματοληψία, με μελέτες όμως που αντιμετωπίζονται με μεγάλη ε, σοβαρότητα και ως εκ τούτου αναμένεται σε ένα σχέδιο δράσης να δοθούν οι λεπτομέρειες που θα οδηγήσουν και στην υλοποίηση και, τα... Ε, και πιο λεπτομερή σχέδια. Σε ευχαριστώ Κάρλο. Όσον αφορά τις δοκιμές σε ζώα. Νομίζω ότι υπάρχει σαφής δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και νομικές απαιτήσεις ε, για την ε, εξάλληψη αυτού που πραγματοποιείται ακόμη ακόμα, διότι δεν έχουμε ακόμη απολύτως κατάλληλες εναλλακτικέ μεθόδους. Ε, παρόλα αυτά, ε, αναπτύσσονται τώρα και μειώνονται οι δοκιμές σε ζώα. Έχουμε την οδηγία για τα ζώα εργαστηρίων και στο πλαίσιο της σχετικής έκθεσης θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. γιατί δεν μπορούμε να ενεργούμε πιο γρήγορα και αναφέρθηκαν οι ενώσεις φθορείου ως παράδειγμα. Μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα σε πολλές περιπτώσεις όμως ε, απαιτείται αρκετός χρόνος για να ληφθεί μια τελική απόφαση διότι πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση, πρέπει να εξεταστεί και η κοινωνική κατάσταση, η οικονομική και άλλες. Ε, και γι' αυτό στον έλεγχο καταλληλότητα έχουμε θίξει το θέμα αυτό και έχουμε υποδείξει ότι εξετάζοντας ε, τις ουσίες σε ομάδες ε, μπορεί να είναι καλύτερη μέθοδος. Το να ομαδοποιούμε λοιπόν ε, τις χημικές ουσίες θα μας επιτρέψει να ενεργούμε πιο γρήγορα και πιο οικονομικά και πιο αποτελεσματικά όσον αφορά την ε, υποκατάσταση για να αντιστραφεί η τάση που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αυτό το έχουμε δει και στο πλαίσιο του REACH. Ε, βλέπουμε μείωση του αριθμού επικίνδυνων χημικών, ωστόσο φαίνεται σαν να αυξάνεται ο αριθμό του επειδή έχει, έχουν ταξινομηθεί πολύ περισσότερες ουσίες ε, στην κατηγορία των ε, επικίνδυνων. Έχουμε όμως μέτρα διαχείρισης κινδύνου και έτσι περιορίζουμε την έκθεση σε αυτές τις επικίνδυνες ουσίες. Έτσι έχει δομηθεί η νομοθεσία περί χημικών και στόχο έχει να μειώσει την ε, έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Ρωτήθηκε γιατί δεν έχουμε περισσότερη δράση τη στιγμή που έχουν εντοπιστεί τόσα προβλήματα στον έλεγχο καταλληλότητας. Ο στόχο του ελέγχου καταλληλότητα ήταν να εξεταστούν πάνω από 40 νομοθετικέ πράξει και να εντοπιστούν τα προβλήματα. Αυτό έγινε, αλλά ε, ο έλεγχο καταλληλότητα δεν υποβάλλει προτάσεις ε, επίλυσης, ε, απλά εντοπίζει τα προβλήματα. Σε επόμενη φάση θα γίνει αυτό και θα γίνει από την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εμεί περιμένουμε εξίσου ανυπόμονα με εσά να δούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό, όπως ε, είπε ο συνάδελφος, δεν μπορούμε να σας πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να περιμένουμε να αναλάβει καθήκοντα η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά το μη τοξικό περιβάλλον και τη σχετική στρατηγική, αυτό αποτελεί απέτηση στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος, το οποίο παρεπιπτόντως ε, θα συνεχίσει να τρέχει μέχρι του χρόνου. Ε, το θέμα της στρατηγικής αυτής όμως είναι ότι σχεδιάστηκε για να αντιμετωπιστούν τέσσερα συγκεκριμένα θέματα τα οποία είναι πολύ επίκαιρα θέματα, πραγματοποιούνται εργασίες και στους τέσσερις τομείς, αλλά όπως ίσως να θυμάστε και από την έλεγχο καταλληλότητα και από την καταλληλότητα και από τον, και από το REACH, ε, έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά τα τέσσερα. Γι' αυτό μάλλον ε, θα χρειαστεί μια πιο ευρία οπτική από την στρατηγική για το μη τοξικό περιβάλλον. Αλλά και πάλι αυτό εναπόκειται στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αποφασίσει. Η κυρία Φόντερ ε, έχει κάνει σχετικές ανακοινώσεις ε, και θα βρείτε και τις σχετικές δράσεις. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Κάρλος σχετικά με την συμμόρφωση με την ομοθεσία REACH. Οι ουσίες που δεν συμμορφώνονται ε, θα υπόκειται σε σχέδιο δράσης το οποίο ήδη έχει συμφωνηθεί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών. Έχουμε εκτελεστική πράξη που προβλέπει ε, κατά τέσσερις φορές αύξηση των ε, ελέγχων των χημικών ε, και θα έχουμε επίσης διευκρίνηση σχετικά με το μέχρι πότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικαιροποιούν τους ε, φακέλου, τα έγγραφα με τα οποία ε, διοχετεύουν στην αγορά τα χημικά. Αυτό λοιπόν θα βελτιώσει την προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τηρήσατε και το χρόνο ομιλία σας. Μας δώσατε μια σειρά απαντήσεων ε, οι οποίες ήταν πολύ σε δεδομένου του χρόνου που είχατε στη διάθεσή σας. Ε, κάποιοι συνάδελφοι όμως μπορεί να θέλουν να επανέλθουν. Ε, έχουμε λοιπόν δύο μιλητές στον επόμενο γύρο. Ε, αν λοιπόν θέλετε κάποια διευκρίνηση στην απάντηση που ακούσατε, παρακαλώ να ζητήσετε το λόγο. Η Μύρια Μταλή. Ναι, Πρόεδρε. Από διαφορετική Τυχή δεν θέλω να το εξετάσω εγώ. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας των χημικών και άλλων κλάδων της βιομηχανίας και ότι εμφανίζονται νέες βιομηχανικές δομές. Ωστόσο, δεν έχουμε αρκετή έμφαση δώσει σε πολιτικές οι οποίες θα διευκολύνουν τις αλλαγές, τις δομές και θα δημιουργήσουν έναν τομέα ο οποίος γνήσια θα δίνει απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις και χρειαζόμαστε ε, μία βιομηχανία χημικών προϊόντων που θα δώσει την όθηση και για καλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και για την αντιμετώπιση της ε, ε, των της στο περιβάλλον και της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να δούμε όμως πώς μπορεί αυτή η νομοθεσία που έχουμε να διευκολύνει και συγκεκριμένα να δώσει όθηση προσλήσεις και για τη βιομηχανία των χημικών και για την ε, γεωργία, προσλήσεις ε, πράσινες, προσλήσεις που θα έχουν, ε, που θα έχουν ουσιαστική συμβολή στην κύκλικη οικονομία. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας και με κάλυψη των αναγκών σε χημικές ουσίες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια σειρά ερωτήσεων, γιατί ήμουν μέλος Επιτροπής για τα ζεσανιοκτώματα στην προηγούμενη βουλευτική περίοδο και ακριβώς εξετάσαμε το θέμα των χημικών ουσιών. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν με έκπληξη διαπιστώνω ότι η ΕΦΣΑ, η Υπηρεσία Ασφάλειας των Τροφίμων, είχε κάνει μια πρόταση για αξιολόγηση των κινδύνων από ζεζαμιοκτώνα για τις μέλισσες, λαμβάνοντας υπόψη ε, και καταμετρώντας την χρονική ε, τοξικότητα των ζεζαμιοκτώνων σε, μια, σε όλη την ηλικία του ζώου, δηλαδή από την, ε, από την ύμφη μέχρι το όριμο έντομο μέχρι τη μέλισσα, που δεν δέχτηκαν όμως τα κράτη-μέλη. Και εδώ ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να το κοιτάξουμε αυτό, γιατί ε, βλέπουμε ήδη να μειώνονται με ραγδαίους ρυθμούς οι αριθμοί των μελισσών. Πρέπει λοιπόν να το προβλέψουμε αυτό. Επίσης, η Santé Publique France, η οποία ε, κάνει αξιολογήσει για τα θέματα αυτά, μας λέει το εξής. Είναι έξι οι ενδοκρινολογικοί διαταράκτες που εμπλέκονται και μπορείτε να διαπιστώστε κι εσείς πως η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είναι επαρκής. Ξέρουμε πως έχουν ε, συνέπειες, τις αντιμετωπίζουν όλοι. Δεν βρίσκονται μόνο στα τρόφιμα ή στα καταναλωτικά αγαθά, βρίσκονται παντού. Το οποίο σημαίνει ότι δεν είμαστε αρκετά αυστηροί στην προσπάθεια απαγόρευσης χρήσης αυτών των ουσιών. Και κάτι ακόμα που μας ανησυχεί και θα θέλαμε εδώ να έχουμε έγκριση από τη σχετική νομοθεσία είναι τα καταναλωτικά αγαθά. Οι πάνες, για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τη βιομηχανία να μας αποκαλύψουν ε, πώς τις ε, παρασκευάζουν, αλλά βρήκαμε ε, κατάλοιπα από εντομοκτώνα, βρήκαμε ενδοκρινολογικούς διαταράκτες. Ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό βρίσκεται όχι μόνο στις πάνες, αλλά και στα αγαθά γυναικείας υγιεινής. Ε, δεν θα έπρεπε να έχουμε σχετική απέτηση για τα σωματίδια αιωρούνται παντού. Στα τρόφιμα βρίσκονται, στα φάρμακα, στα εμβόλια. Και δεν γνωρίζουμε τίποτα για τα σωματίδια αυτά. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει πως χρειάζεται και σχετική νομοθεσία. Είτε να φτιάξουμε λοιπόν ένα ρίτς για τα νάνο σωματίδια, γιατί όταν περάσαμε από τη Σχετική Επιτροπή ρίτς, καταλάβαμε πως είναι. γίνεται καταχώρηση μέσω ριτς και η ε, βιομηχανία φρόντιζε να φύγουν από την κυκλοφορία, ακόμα και αν ο φάκελο, με συγχωρείτε, έβγαιναν στην κυκλοφορία, ακόμα και αν ο φάκελο δεν ήταν πλήρη. Από εδώ και πέρα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Θα πρέπει να είναι πλήρη ο φάκελο πριν κυκλοφορήσουν. Έχουμε τεράστια κενά στο σύστημα, γιατί παρά είστε καλοί με τους βιομηχανικούς κύκλους. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Και πιστεύω πως και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο ισχύει το ίδιο. Δεν είμαστε αρκετά δυναμικοί. Δεν δείχνουμε πυγμή όταν μιλάμε για το περιβάλλον. Όλοι αργοπαθαίνουμε από καρκίνους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το Προεδρείο που έβαλε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ όσου πήραν το λόγο και τι εξηγήσει που δώσανε. Έχω λοιπόν μία παρατήρηση που ενδεχομένω σα φανεί προκλητική. Αναφερθήκατε στι ανησυχίε σα για του δισταγμού των βιομηχανικών κύκλων, για τα όσα μίλησε ο κύριο Ριβαζή και επίση είπατε πω ανησυχείτε για τι διάφορε πρωτοβουλίε τη μεμονωμένη των κρατών μελών. Όταν λοιπόν αναφέρεστε σε όσου δέχονται του κανόνε, ποιοι είναι οι κυβερνήσεις, η βιομηχανική κλάδη και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιοι άλλοι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορούν ε, είτε μέσω μπλε κάρτας να πιέσουν ε, τους κύκλους αυτούς, είτε τις κυβερνήσεις. Οι πολίτες μας, γιατί η νομοθεσία μπορεί να έχει μία διετή προσέγγιση που είναι έγκριση και ε, αδειοδότηση, αλλά μπορεί να βασίζεται και στην ενημέρωση των βασικών εμπλεκομένων που είναι οι καταναλωτές και ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες συνηγορούν υπέρ ενός συστήματος ε, σήμανσης, μα όπως το Nutri-Score ε, για τα διατροφικά, το οποίο χρησιμοποιούν ευρύτατα και το οποίο επιτρέπει να έχει κανείς την ενημέρωση που χρειάζεται ως κοινό για τα προϊόντα που χρησιμοποιεί. Η ερώτηση μου είναι το εξή. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές είναι αρκετά ενημερωμένοι για αυτές τις νομοθετικές προσεγγίσεις για να τις ε, χρησιμοποιήσουν. Και δεύτερον, θα χρησιμοποιήσετε εσείς τη δυνατότητα ενημέρωσης με κατάλογο ε, ουσιών και με βαθμολογία έτσι ώστε τα πράγματα να βελτιωθούν. Έχουμε τρεις ε, ομιλητές που έκαναν ερωτήσεις. Ε, θα πρότεινα οι ερωτήσεις να είναι σύντομες, έτσι ώστε οι συνάδελφοι ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσουν να απαντήσουν. Θα είμαι πολύ σύντομη. Διαδικασία fast track όταν διαπιστώνουμε πως υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες. Εσείς θα συστήσετε σε εμά να ακολουθήσουμε μια διαδικασία fast track όταν διαπιστώνουμε τέτοιου είδους ουσίες μεμονωμένα. Αυτό θα ήταν καλό γιατί θα μας επέτρεπε να αλλάξουμε μια ολόκληρη γκάμα νομοθεσία. Δεύτερον, το μήνυμα δεν είμαι σίγουρη το κατάλαβα. Θα επιτρέψετε ή όχι στην κυβέρνηση της Δανίας να ε, ε, απαγορεύσει κάποια από, αυτές, κάποια από αυτά τα συστατικά ε, σε υλικά ε, επαφής με τρόφιμα τα οποία μεταναστεύουν στο ίδιο το τρόφιμα και το οποίο η Δανία επιθυμεί να απαγορεύσει. Γιατί δεν κατάλαβαν η απάντηση σας στην αρνητική ή η θετική. Ε, και εμένα η ερώτηση μου είναι πάρα πολύ σύντομη. Θέλω να επιμείνω στη στρατηγική για το μη τοξικό περιβάλλον που έχει περιγραφεί στο έβδομο ε, σχέδιο για το περιβάλλον ως νομική υποχρέωση. Καθυστερείται και δεν καταλαβαίνω πώς η καθυστέρηση αυτή θα μας βοηθήσει στο να εξασφαλίσουμε πώς το περιβάλλον αυτό θα το ε, εξασφαλίσουμε και για τους ανθρώπους, όχι μόνο για τη βιοπικιλότητα. Επίσης, έχουν γίνει παρατεταμένες συζητήσεις για το REACH που δεν είναι το θέμα σήμερα. Και για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έθιξα, σας ρώτησα δράση, όχι λόγια. Θα δούμε τι θα κάνει η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τέσσερα χρόνια εσείς εξετάζετε όλα αυτά και ε, τις ε, ασυνέπειες στην αξιολόγηση κινδύνων, στους διαταράκτες, στην σόρευση και δεν έχετε καταθέσει καμία πρόταση. Και δεν ξέρω πώς να το πω χωρίς να γίνω αγενής αλλά εν πάση η προσδοκία μου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να κάνει τη δουλειά της. Um, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις που έδωσε, αλλά παρόλα αυτά είστε ασαφείς. Θα ήθελα να μου δώσετε μία απάντηση για το γενικότερο θέμα που μας ε, ε απασχολεί, που είναι το χρώμιο 6. Εκεί έχουμε βασικό πρόβλημα, γιατί ο γεωμηχανικός κλάδος θεωρεί και τα λόμπι τους πως δεν χρειάζεται νομοθεσία. Η πολιτική ε, έχουν ε, διαφορετικές γνώμες, κάποιοι είναι πιο ανοιχτοί στο λόμπινγκ ή όχι και για το λόγο αυτό είναι ουσιαστικό να δώσουμε το λόγο στον επιστημονικό κόσμο, στους ανεξάρτητους επιστήμονες και να μην ακούμε πια αυτούς οι οποίοι για λόγους προσωπικούς, πολιτικούς, οικονομικούς γέρνουν προς τη μία ε, ή την άλλη κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή ευρωπαικη επιτροπη για το θέμα αυτό συμφωνείτε για, το, για την έκθεση της Επιτροπής για τα ζακνιοκτώνα και όταν μιλάμε για το ρίφιτ θα αλλάξει κατα κατάσταση ριζικά. Ποιε είναι οι προθέσει σα και αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ, Γιούτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους. Κάποιε από τις απαντήσεις δεν ήταν αρκετά σαφείς λόγω της ε, και σοβαρής κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Επαναλαμβάνω, όχι μόνο τα όσα είπαν οι συνάδελφοι, εμείς χρειαζόμαστε να δούμε αυτή τη στρατηγική πια που τόσο καιρό περιμένουμε για το μη τοξικό περιβάλλον. Τόσο καιρό πια περιμένουμε. Τόσο καιρό έχετε καθυστερήσει. Μα δεν είναι σοβαρό να μην ε, την παρουσιάζετε. Και θα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι εμείς λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά το θέμα του περιβάλλοντος και της προστασίας της υγείας τους. Και επίσης θέλω να τονίσω πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση με τους ενδοξινολογικούς διαταράκτες. Έχουμε τις μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει σύνδεση με σοβαρές ασθένειες και προβλήματα γονιμότητας στα κράτη-μέλη. Και πρόσφατα συναντήθηκα με καθηγητή που συζήτησε την κατάσταση κάνοντας μια μελέτη σε έγκυες γυναίκες και ε, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ε, βρήκαν να έχουν ε, ε, στις αναλύσεις υψηλά επίπεδα ενδοκρινολογικών διαταρακτών, κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία του μωρού όταν γεννιέται. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο σύνδεσμος και πρέπει να τα καταφέρουμε όλα αυτά για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και τις μελλοντικές γενιές. Θα λογοδοτήσουμε για το θέμα αυτό. Προστατεύσαμε τα νεογέννητα ή όχι. Δεν θέλουμε ενδοκρινολογικούς διαταράκτες μόνο για ένα πληθυσμιακό, μια πληθυσμική ομάδα. Όχι, παντού. Πόσιμα, καλλιντικά, ε, πλαστικά, παντού. Τι θα κάνετε λοιπόν για τους ενδρολικούς διαταράκτες. Ποια θα είναι η δράση σας. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Ακούσατε λοιπόν πως οι συνάδελφοι ανησυχούν πολύ είναι ένα θέμα βασικής ε, εμπιστοσύνης των πολιτών στα προϊόντα τα οποία αγοράζουν και στα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουν, όπως επίσης και στο νερό το οποίο πίνουν. Τι έκθεση έχουν ε, σε χημικά στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Σας παρακαλώ πολύ, απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις και καταλαβαίνω ότι ο χρόνος δεν υπάρχει, καταλαβαίνω τις δυσκολίες, καταλαβαίνω πως έχετε δώσει αρκετά συγκεκριμένες απαντήσεις πριν, αλλά το τονίζω. Αν οι συνάδελφοι φύγουν από τη συνάντησή μας με την αίσθηση ε, πως ακόμα έχουμε ε, ασάφειες, δεν θέλουμε να περιμένουμε μέχρι τη νέα θητεία της Επιτροπής, θέλουμε η δράση να αναλυθεί τώρα. Yes, thanks. Ναι, σας ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να είμαστε σαφείς. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι αυτή τη στιγμή έχει εκλεγεί μόνο η πρόεδρος. Και στις γενικές κατευθυντήρες γραμμές της παίζουν σημαντικό ρόλο η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία της υγείας των πολιτών. Όχι μόνο το κλίμα αποτελεί προτεραιότητα, αλλά και το περιβάλλον. Και υπάρχουν και άλλα κεφάλαια, όπως είναι η προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και η προστασία των ανθρώπων. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στις κατευθυντικές γραμμές, αλλά αποτελούν απλά κατευθυντικές γραμμές. Δεν είναι πρόγραμμα εργασίας. Για να γνωρίζουμε λοιπόν τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει πρώτα να οριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν θα αναλάβει τα καθήκοντά τη, ελπίζουμε την 1η Νοεμβρίου. Και κατόπιν θα μπορέσουμε να λάβουμε αποφάσει και να δεσμευτούμε. Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να πούμε τι ακριβώ θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη στιγμή που δεν ξέρουμε καν ποια θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόγραμμα εργασία. Θα προσπαθήσω πάντω να σα δώσω περισσότερε διευκρινήσει πάνω σε κάποιε ερωτήσει. Στην κυρία Νταλή να πω σχετικά με τη βιομηχανία ότι απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν ε, στον τομέα αυτών της οικονομίας, ε, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια δουλειά τα τελευταία πέντε χρόνια. Πριν πέντε χρόνια υπήρχε, ε, υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήξεραν τι είναι η κυκλική οικονομία. Ε, σήμερα μιλάμε όλοι για τα, για τα πλαστικά Έχουμε ε, νομοθεσία, ε, έχουμε μια πρωτοβουλία, ε, έχουμε απαγόρευση για τα πλαστικά μίας χρήσης που αποτελούν από τα σημαντικά προβλήματα για το περιβάλλον και τώρα πια δεν θα αποτελούν απόβλητα αλλά θα αποτελούν δευτερεύοντα υλικά. Έχει έχει γίνει λοιπόν ε, πολλή δουλειά, αλλά δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα μέσα σε πέντε χρόνια. Πρόκειται λοιπόν για μια προτεραιότητα που συμπεριλαμβάνεται στις κατευθυντήρες γραμμές ε, της ε, νεοεκλεγής σας Προέδρου. Το να συνεχιστούν δηλαδή οι εργασίες πάνω στην κυκλική οικονομία. Όσον αφορά τη πολύ συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με ε, το χαρτί ψησίματος ε, στην Δανία. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κοινοποίηση από τη Δανία που να ζητάει παρέκκληση, αλλά Έχουμε εκατοντάδες τέτοιες ε, υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Τη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως δεν την γνωρίζω. Και τώρα θα περάσω στην ερώτηση που διατυπώθηκε στα γαλλικά για την σήμανση των ε, περιβαλλοντικών προϊόντων και θα ήθελα να πω ότι έχουμε πολύ λεπτομερή σήμανση και από τις πιο προηγμένες του κόσμου στην Ευρώπη, αλλά χρειάζεται μια συνθετική προσέγγιση. Έχουν ε, πραγματοποιηθεί μελέτες από τους αδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι εκείνη η οποία θα μπορέσει να κάνει τις προτάσεις της, τις νομοθετικές προτάσεις. με τη νέα τη σύνθεση, αλλά και χωρίς να μπορώ να προβλέψω τις αποφάσεις που θα ληφθούν αργότερα, καθώς έχει γίνει πολλή δουλειά μέχρι τώρα, φαντάζομαι ότι η νέα Επιτροπή θα συνεχίσει πάνω στην ίδια γραμμή. Και τώρα θα μου το δόλος, να δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Και θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω στην ερώτηση σχετική με τα απόβλητα που ακούστηκε νωρίτερα. Νέα νομοθεσία για την ταξινόμηση των αποβλήτων και τους νέους ορισμούς ε, τέθησε ισχύ πέρσι, αλλά πρέπει ακόμα να υλοποιηθεί από τα κράτη-μέλη, όπως και γίνει αυτό, θα είναι πιο σαφής η κατάσταση για το τι συνιστά απόβλητο και τι όχι. Ε, πρέπει να τηρηθεί λοιπόν αυτή η νέα νομοθεσία είναι νέος νόμος και άρα ακόμα δεν έχει μεταφερθεί από τα κράτη-μέλη. Αυτό πρέπει να παρακολουθήσουμε. Βέβαια, ακόμα χρονικό περιθώριο υπάρχει, δεν έχει λήξει προθεσμία. Για το αν η Επιτροπή είναι επίοικης ή όχι σε σχέση με το πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού των μελισσών και τους επικονιαστές. Θα παρακαλούσα αυτή την ερώτηση να την απευθύνετε στους αδέλφους της αρμόδιας υπηρεσίας γιατί όντως διαπιστώνουν με ανησυχία τη μείωση των επικονιαστών στην Ευρώπη και συμφωνούμε οπωσδήποτε ότι πρέπει να αναλυφθεί δράση στο τομέα αυτών, το δέχετερο δυνατό. Τέλει, μάλλον δύο ερωτήσεις, να υλικά που ανέφερε η κυρία Ριβαζή. Η αλλαγή στις ε, προϋποθέσεις έχει τεθεί σε εφαρμογή σε σχέση με την ε, καταχώρηση υπό τον κανονισμό REACH των νανό υλικών. Με βάση αυτή την καταχώρηση θα γίνεται και η ανάλυση της επικινδυνότητας για το περιβάλλον αυτών των ουσιών και η διαχείριση του κινδύνου για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Αυτά αναφέρθηκαν άλλωστε και από την ε, κυρία Φοντερ Λάιεν ως τομείς δράσης. Η Επιτροπή στην τρέχουσα τη σύνθεση έχει οθετήσει στρατηγική για τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες ήδη από πέρσι. Με πρώτο και κύριο βήμα την επισκόπηση της νομοθεσίας ε, οριζοντίως για το αν υπάρχει επάρκεια νομοθετική, αν χρειάζεται κάποια νομοθετική παρέμβαση, αν ε, μπορεί να φέρει αποτελέσματα μια νέα νομοθεσία, αλλά πρέπει να δούμε πρώτα αυτή την επισκόπηση, να δούμε τα αποτελέσματά της. Και μετά θα υπάρξει και μια πλατφόρμα ε, ως μονοθυριδική προσέγγιση ώστε να μπορεί κανείς όλες τις ε, επιλογές του να τις ε, βλέπει μέσα σε ένα σημείο, σε έναν ιστότοπο. Και έτσι θα έχουμε ουσιαστικές αλλαγές μετά το fitness check αυτό, αυτή την επισκόπηση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις σας. Σημειώνουμε τις ε, υποσχέσεις και δεσμεύσεις της κυρίας Φοντερ Λάιεν βεβαίως και επιμένουμε στις ανησυχίες που διατυπώσαμε και την επιμονή μας να παρακολουθήσουμε εκ του συνεγγύς της περαιτέρω δράσης Επιτροπής Πάντα βέβαια όταν βρισκόμαστε από τη μια σύνθεση επιτροπής ε, μέχρι την ανάληψη καθηκόντων ε, από τη νέα, βλέπουμε η απερχόμενη επιτροπή να διστάζει να λάβει δράση και πολλές φορές ε, να μην υλοποιούνται δράσεις, να μην γίνονται αξιολογήσεις, παρά όταν έχει πια περάσει αρκετός καιρός και έχει έτσι έρθει να οριμάσει το θέμα στους κόλπους της νέας Επιτροπής. Ε, ελπίζω λοιπόν να μην χαθούν τα σημαντικά θέματα που μας απασχολούν και που γύρουμε εδώ στις, ε, στην εναλλαγή αυτή σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε και για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Thank you, the Ανταλλαγή με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 07-2019 πρόκειται για μια δράση για ε, την προσφορά υπηρεσίας διασυνοριακής. Ο κύριος Wells στον τομέα του οι συναδέλφοι βεβαίως έχουν το λόγο στη συνέχεια για να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Αν χρειαστεί εγώ να αποχωρήσω χωρίς πρόβλημα οι συνάδελφοι θα με ρημνήσουν. Αλλά το λόγο έχετε το λόγο κύριε Βολής. Ε, thank you very much. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ την ε, ομάδα που εργάστηκε πάνω σε αυτό το θέμα, διότι νομίζω ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι συνεργάστηκε πολύ επικοδομητικά και επαγγελματικά μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ακόμα και σε στιγμές που δεν ήμασταν απόλυτα πεπισμένοι από τις δράσεις που είχαν αναλάβει. Νομίζω ότι έκαναν εξαιρετική δουλειά όσον αφορά τη συνεργασία μαζί μας. go around. Good. Uh, this is, uh, as it's a uh, relatively new parliament, it's just a reminder of the, of the role of, of the Euro. Επειδή ε, τώρα ξεκινάει η θητεία, ήθελα να σας θυμίσω λίγο το ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου, ελέγχει τους ε, λογαριασμούς, ε, υποβάλλει γνωμοδοτήσεις, εγώ θα ήθελα να θίξω ιδιαίτερα το τελευταίο θέμα που είναι η αποτελεσματική χρήση φυσικών πόρων. Με πολύ ενδιαφέρον ακούσαμε τη συζήτησή σας ε, και φέτος ε, είχαμε εκπονήσει είχαμε έκθεση συγγνώμη, ε, για το περιβάλλον ε, και για τα φυτοφάρμακα, κάτι που νομίζω ότι θα ενδιαφέρει και τη δική σας Επιτροπή. Εγώ θα επιστρέψω αργότερα με συναδέρφους για να ακούσουμε τον Επίτροπο Βέλα. μας ενδιαφέρουν γενικά οι εργασίες της Επιτροπής σας και ελπίζουμε και η δική μας δουλειά να είναι χρήσιμη για σας. Η έκθεση αυτή εξέτασε έναν τομέα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι πολύ φιλόδοξες. Έχουμε κάποια δύσκολα θέματα. Εξετάσαμε την εφαρμογή της ε, ε, οδηγίας για την διασυνοριακή περίθαλψη Εξετάσαμε και ε, τις ε, διασυνοριακές ανταλλαγές δεδομένων, κάτι που γίνεται εδώ και 12 χρόνια που αναφέρεται και στην οδηγία και εξετάζουμε και το θέμα των ε, σπάνιων ασθενειών, κάτι το οποίο μας αποσχολεί εδώ και 10 χρόνια συνολικά. Αυτό το διάγραμμα μάλλον είναι δύσκολο να το διαβάσετε αλλά θέλω να σας δώσω μια εικόνα του πόσο πολύπλοκο είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Εδώ βλέπετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούμε να το παρουσιάσουμε τις ε, μετακινήσεις ασθενών ε, σύμφωνα με την οδηγία. Τα... Από τη Γαλλία προέρχονται τα 2% ε, των ασθενών έχουμε τα περισσότερα στοιχεία. Ε, κάνα δύο κράτη-μέλη δεν μας έχουν υποβάλει στοιχεία. Βλέπετε όμως αρκετά πολύπλοκες μετακινήσεις. Βλέπετε κάποιες διμερείς μετακινήσεις, είναι όμως δύσκολο το θέμα αυτό όσον αφορά τις διαδικασίες, αλλά νομίζω κυρίως όσον αφορά τα θέματα πληροφορικής. Εξετάσαμε την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όσον αφορά την οδηγία και εξετάσαμε και τις πρωτοβουλίες για τις ε, σπάνιες ε, ασθένειες όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς και η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα. Εξετάσαμε επίσης τις ανταλλαγές δεδομένων. Εδώ βλέπετε λοιπόν μια επισκόπηση των όσων βρήκαμε. Θα τα διατρέξω αυτά αρκετά γρήγορα. Αν ε, ήταν πιο φιλόδοξη η παρουσίασή μου, ε, θα μπορούσα να ε, έχω βάλει ένα πολύ έντονο πράσινο σημάδι στο πρώτο σημείο ότι τα καταφέραμε, κάπως λιγότερο όμως στα σημεία 2 και 3. Τι βρήκαμε πληροφόρηση των ασθενών όσον αφορά τα δικαιώματά τους για διασυνορική περίθαλψη. Από τότε που ε, τέθηκε σε ισχύ η οδηγία, είναι ατελής ή ασαφής ε, σύμφωνα με κάποιες αναφορές. Φέτος ε, τον Φεβρουάριο το Κοινοβούλιο ε, ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι η πολυπλοκότητα του πλαισίου ε, κάνει πολύ δύσκολο το να εξηγήσει κανείς στους ασθενείς τα δικαιώματά τους και τους κανόνες που ισχύουν για αυτούς. Εμπειρογνώμονες θεώρησαν ότι τα εθνικά σημεία επαφής μπορούν να δίνουν πολύ καλύτερη ενημέρωση στους πολίτες και όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες και αυτό είναι κάτι που αντικατοπτρίζεται στην έκθεσή μας. Οι συστάσεις μας εδώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να υποστηρίξει τις εργασίες των Εθνικών Σημείων Επαφής. Είχαμε την εργαλειοθήκη του 2018 που πιστεύουμε ότι αποτέλεσε θετική εξέλιξη για να γίνουν πιο φιλικά προς το χρήστη τα εθνικά σημεία επαφής. Θα θέλαμε όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει την χρήση των εθνικών σημείων επαφής και πιστεύουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις αναφορές εμπειρογνωμόνων ότι το ε, ευρωπαϊκό δίκτυο θα πρέπει να καλύπτεται από τα εθνικά σημεία επαφής και ε, να παρέχονται ε, σχετικές ε, οδηγίες στους ασθενείς. Όσον αφορά το δεύτερο σημείο που είναι η διασυνοριακή ανταλλαγή ε, δεδομένων των ασθενών, ε, θα ήθελα να εκφράσω την κατανόησή μου για τη δύσκολη θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι είναι πολύ δύσκολο να το κάνει κανείς σωστά αυτό και απαιτεί ε, διαχείριση του προγράμματος ε, πολύ προηγμένη. Όταν ολοκληρώσαμε την έκθεσή μας ε, και νομίζω ότι ακόμα και τώρα η ανταλλαγή δεδομένων με βάση αυτή την αρχιτεκτονική γίνεται σωστά μόνο από την Φιλανδία προς την Εστονία. Η ευρύτερη χρήση λοιπόν της αρχιτεκτονικής αυτής ε, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Πολλά κράτη-μέλη είναι έτοιμα να λάβουν δεδομένα, αλλά δεν δεν υπήρχαν πολλά κράτη-μέλη όταν εμείς ολοκλώσαμε τον έλεγχό μας που να είναι έτοιμα να στείλουν δεδομένα. Δεν ήταν λοιπόν τόσο επιτυχές αυτό το εγχείρημα όσο ελπίζαμε αρχικά. Και θεωρήσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν μάλλον αρκετά φιλόδοξη όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό και ήταν αρκετά ε, αισιόδοξη, δεν καταλάβαινε πόσο δύσκολη θα ήταν η εφαρμογή του. Για να έχουμε καλύτερες ε, διασυνοριακές ανταλλαγές ε, δεδομένων στο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρήσιμο θα είναι να διενεργήσει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση των ε, όσων έχει κάνει μέχρι τώρα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιες ε, διμερείς ρυθμίσεις ανάμεσα σε κάποια κράτη-μέλη, υπάρχουν δηλαδή κάποιες διμερείς ροές, ε, αυτό μάλλον είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσω στο πολύ δύσκολο και φορτισμένο θέμα των σπάνιων ασθενειών. Νομίζω ότι όλοι μας θα θέλαμε να δούμε σημαντική πρόοδο στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2008 ε, έχει σχετική προσέγγιση και από το 2014 είχαμε κυρίως ε, τα ERN ε, που όμως αποτελούν σημαντική πρόκληση για την ε, οικονομική βιωσιμότητα. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δίκτυα και η αξιολόγηση της ε, δουλειάς των εταίρων ε, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο θα είναι το μέλλον αυτών των δικτύων, των ERN, των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς. Το πλαίσιο ίσως ε, να μην είναι αρκετά σαφές ε, και δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Τι αναζητούμε λοιπόν. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναξιολογήσει τη στρατηγική της, ε, να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλη ή αν θα πρέπει να τροποποιηθεί ελαφρά ή σε σημαντικό βαθμό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περιγράψει τρόπους να αξιολογηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δίκτυα και εάν τα δίκτυα είναι να συνεχίσουν η υπομορφή παρόμοια με τη σημερινή, θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με τη διαφάνειά τους. Συνοψίζοντας λοιπόν, ε, παρατηρούμε πρόοδο σε κάποιους τομείς όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. Απομένουν πολλά να γίνουν, ε, μεταξύ άλλων ε, αξιολόγηση των όσων έχουν γίνει και αξιολόγηση των τρόπων που προτείνεται να προχωρήσουμε. Το Κοινοβούλιο έχει ένα έγγραφο του Φεβρουαρίου για το θέμα αυτό και συμφωνώ με τα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου ότι μια τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει η υπόψη ε, το, τις συνέπειες ως προς την ε, ποιότητα ζωής των ασθενών. Ελπίζω τα, η δουλειά που κάναμε εμείς να αποτελέσει σημαντική και επικοδομητική συμβολή στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε Βόλκερ, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ και για την παρουσίαση. Η έκθεση εφαρμογής Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει επαρκώς. Και αυτό το καταγράφει και το ελεκτικό συνέδριο. Μπορεί να έχουμε φιλόδοξα μέτρα να έχει εισαγάγει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλόδοξα μέτρα, αλλά δεν επετέφθησαν οι στόχοι σε πολλές περιπτώσεις και πολύ συχνά ιδιαίτερα η διαχείριση των αναγκών και των ωφελών για τον ασθενή πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά και είπατε και εσείς ότι μιλούμε για την διάρκεια, για την αηφορία στην ικανοποίηση των αλλαγών οι πολίτες λοιπόν δεν ενημερώνονται παρκώς για τα δικαιώματά τους. Δεν βλέπουμε όφελος από την κάλυψη, τη διασυνοριακή. Μας είπατε άλλωστε και εσείς ότι μόνο ένα κράτος έχει, ε, κάνει, έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα. Θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ο ψηφιακός τομέας είναι, πιστεύω, σε μεγάλη καθυστέρηση, ενώ έχει τεράστιο δυναμικό, δεν το έχει αναπτύξει. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσίαση και συμφωνώ με τις συστάσεις σας η, Ευρω... η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πιστεύω να τις ακολουθήσει, θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία. Σας ευχαριστώ και πάλι. Um, ε, good morning. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας παρουσιάσατε. Έχω τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν πιστεύω πολύ πως θα πρέπει να στήσουμε εξειδικευμένα κέντρα για τις σπάνιες ασθένειες στην Ευρώπη, τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένα στο δίκτυο αναφορών. Θα ήθελα πολύ να καταλάβω ποια είναι τα πραγματικά εμπόδια τα οποία εξηγούν αυτή την πολύ αργή ε, παράδοση αυτών των κέντρων, ε, σύμφωνα με το όσοι εσείς ξέρετε. Λυπάμαι πολύ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο συστήματα ε, που δρούν παράλληλα. Πώς θα δώσουμε λοιπόν ε, περισσότερη ενημέρωση. Υπάρχουν τα εθνικά σημεία επαφής, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε πολλές προσπάθειες για την ενημέρωση, για την πρόσβαση στα φάρμακα, στις, ε, ιατρικές, ε, στην ιατρική περίθαλψη, στις θεραπείες, σε όλους τους πολίτες για να έχουν την ίση ευκαιρία στη διάγνωση, στη θεραπεία, στην ποιότητα ζωής κάποια κράτη-μέλη περιμένουν στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουν πιο σαφείς κανόνες για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για την παραπομπή ασθενών. Για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το πώς θα στηρίζονται από το κράτη-μέλη ε, και πώς θα στηρίζουν τα κράτη-μέλη το δίκτυο, σας ρωτώ το εξής χρειάζεται αύξηση της στήριξης από τη δική σας πλευρά. Έχω και άλλες ερωτήσεις, θα τις αφήσω για αργότερα και δι... ελπίζω ε, οι συνάδελφοι να κάνουν τις υπόλοιπε ερωτήσεις. Ευχαριστώ ε, η συνάδελφο. Σας ευχαριστώ και εγώ για το θέμα των διασυνοριακών, τη διασυνοριακής περίθαλψης. Φιλόδοξα μεν, αλλά καθυστερημένα. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Ένα από το πρόβλημα στην εφαρμογή και έχει ακουστεί προηγουμένως είναι το πώς συγκεκριμένο ε, πώς συγκεκριμένα θα γίνεται αυτή η ενημέρωση από τα κρατη γιατί δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη μέρος του δικτύου, δεν έχουν όλοι συστήματα περίθαλψης online, άρα λοιπόν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών οι πολίτε είναι απαραίτητο να έχουν αυτές τις πληροφορίες και να ενημερώνονται, για παράδειγμα, για τιμή φαρμάτων, για κάλυψη, ε, για αποζημίωση, για ε, θεραπείες και κυρίως για ασθενείς που ε, υποφέρουν από σπάνιες ασθένειες για τις οποίες δεν πρέπει κανείς να καθυστερεί τη θεραπεία. Χρειάζεται λοιπόν μία απόφαση εσείς πιστεύετε πως χρειάζεται ένα προστατευμένο ε, πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου θα γίνεται η ενημέρωση για την τιμή των φαρμάκων σε κάθε κρατημέλη που θα έχουν πρόσβαση όλες οι διοικήσεις οι σχετικές των κρατών μελών έτσι ώστε να γνωρίζουν τι γίνεται. Θεωρείτε πως η τρέχουσα οδηγία επιτρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συνεισφέρει κατά την άποψή σας. Στηρίζουν κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να το πω με ταπεινότητα παρουσιασμένη ε, κατάσταση. Αυτές οι σπάνιες ασθένειες και το δίκτυο το σχετικό είναι ένας χαρακτηριστικός κλάδος που είναι απαραίτητη η ευρωπαϊκή παρουσία για τον ασθενή. Είμαι ογκολόγος στην Γαλλία και έχουμε κάποιους σπάνιους ε, καρκίνους, για παράδειγμα παιδικούς καρκίνους που τα χρειάζονται. Και γι' αυτό είναι ανησυχητικό για μένα όταν δηλώνεται πως το μέλλον αυτού του δικτύου ίσως τεθεί υποσφυδίτηση. Και θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτές οι αμφισβητήσεις. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ το λεκτικό συνέδριο για την έκθεση. Ένα ζήτημα που με ανησυχεί ιδιαίτερα ήθελα να θίξω. Βλέπουμε από τα δεδομένα της Eurostat ότι 2,9 των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ηλικία ε, σε ενεργ, του ενεργού πληθυσμού ε, διέμενε σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ένα πολύ μικρό ποστό κάτω από το 0,5% αξιοποίησε τις δυνατότητες που προσφέρει η οδηγία για τις διασυνοριακές ε, υπηρεσίες υγείας. Άρα το σύστημα δεν ε, ωφελεί, του μάλιστα αποθαρρύνει τον ε, πολίτη όταν μένει σε άλλο κράτος μέλος. Και ρωτώ εάν έχει αναλυθεί αυτός ο παράγων από το ελεγκτικό συνέδριο για την προετοιμασία της έκθεσης. Ευχαριστώ κύριε Ριβαζή. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Έχω μια πρώτη ερώτηση. Όταν μας παρουσιάσατε αυτή την διαφάνεια, μας δείχνατε ροές από τη μια χώρα στην άλλη. Μου εξηγείτε λίγο τι ροές είναι αυτές. Δηλαδή αυτοί που, έχουν, που ξεκινάνε από τη Σουηδία για την Ορβηγία, γιατί να πάνε στην Ισπανία, λόγω τιμή, λόγω κόστους, επειδή είναι καλύτερα τα νοσοκομεία ή γιατί είναι σταξιούχοι και καθίστανται εκεί στην Ισπανία για τη σταξία του. Θέλω κάποιε εξηγήσει. Και για τη Γαλλία δεν μας πάτε τίποτα. Είναι γιατί δεν σας έδωσε στοιχεία η Γαλλία. Ναι, μια εξήγηση στο. Επίση, στι ε, θεραπείες και αγωγές. Η νόσος του Λάιμε, παραδείγματι, βλέπουμε. Πολύ, ξέρω ότι πολλοί Γάλλοι πάνε στη Γερμανία γιατί ήταν διαφορετικές οι διαγνώσεις που, είχαν, που μπορούσαν να λάβουν. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, ε, όπως ε, το Λεβεροτιρόξ ως ε, φάρμακο που είχε γεννήσει προβλήματα στη Γαλλία αντικαταστάθηκε από ένα άλλο συναφές που αναζητούσε ο ασθενής στη Βέλγιο, τη Γερμανία κτλ. Άρα και σε αυτό υπάρχουν κάποιες ε, ροές που πρέπει να εξηγηθούν. Επίσης στη Γαλλία έχουμε ελλείψεις φαρμάκων γιατί υπάρχουν αφενός με ομαδικές αγορές ε, όμιλοι συγγνώμη, αγορών ε, στις, ε, από φαρμακεία που προτιμούν να πωλήσουν σε χώρες του εξωτερικού που θα είναι πιο υψηλή, υψηλή η τιμή που θα μπορέσουν να πάρουν και επίσης ε, γιατί η φαρμακοβιομηχανία δεν παράγει προϊόντα όταν αυτά βγαίνουν εκτός της προστασίας ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, γιατί δεν τη συμφέρει. Έχετε λοιπόν κάποιες ε, εντοπίσει κάποια ζητήματα εδώ και μπορείτε να προτείνετε κάτι. Υπάρχει παραδείγματι μια ιδέα, όπως βλέπουμε στις ΗΠΑ, ότι παράγονται φάρμακα ε, πρώτης ανάγκης και μάλιστα και ενεργές ουσίες. Γιατί τώρα πολύ μεγάλο ποσοστό των αργών ουσιών προέρχεται από την Ασία, παράγεται στην Ασία και άρα δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις πρώτες ανάγκες, τις πρωτορχικές ανάγκες των ασθενών εφόσον αυτά τα φάρμακα δεν παράγονται σε ευρωπαϊκά κράτη. Μήπως λοιπόν ο, η λύση θα ήταν, γιατί βέβαια οι ιδιωτικέ εταιρείε δεν έχουν τα ίδια μελήματα με τις δημόσιες, να ε, καθιδρυθεί ένας, να θεσπιστεί ένας δημόσιος φορέας που θα παράγει τα φάρμακα αυτά και τις ενεργές ουσίες, τις δραστικές ουσίες. Ευχαριστώ. Κυρία Κουσένσικα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ε, πολύ αξιόλογη δουλειά που κάνατε. Και θα ήθελα να μου πείτε οι διατάξεις αυτές, σε πώς μπορούν να υλοποιηθούν. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει α, τις ε, την κάλυψη την υγειονομική. Έχει προσφερθεί κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να δράσουμε κατά τρόπο εναρμονισμένο, ώστε να προσφέρεται στον πολίτη ικανοποιητική τεχνολογία, ε, ικανοποιητική υπηρεσία και τεχνολογία στην υγεία. Δεν πρέπει να γίνει μια καταγραφή των υπηρεσιών που προσφέρονται διασυνοριακά. Γιατί αυτή η υποστήριξη ε, είναι όρος που θα κρίνει και την ποιότητα της δημόσιας υγείας. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές, σε παραδείγματι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά το μέλλον, δεν έχουμε δηλαδή ακόμα ουσιαστικές ε, λύσεις. Κι όμως η σύγχρονη τεχνολογία είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί καλή υπηρεσία που θα προσφέρεται διασυνοριακά στον πολίτη όταν ταξιδεύει ηλεκτρονικά. Ένα απλό παράδειγμα, το ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό ενός πολίτη που θα πρέπει να είναι προσβάσιμο όταν ταξιδεύει σε μια άλλη χώρα ή σπάνιες ασθένειες που μπορούν να δώσουν στοιχεία σε όρους big data πολύ πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρηματοδότηση λοιπόν, τι προβλέπετε να γίνει για αυτήν, πώς μπορούν να συνταθούν μεταξύ τους τα εθνικά συστήματα. Και βέβαια αυτό το ρωτώ ε, έχοντας γνώση και των σημαντικών πολιτικών δυσκολιών Μύρια, με συγχωρείς, παρότι είχα δει, δεν σημείωσα το όνομά σου και σε ξέχασα. Μα και εγώ νόμιζα ότι με αγνοείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Θέλω να επαναλάβω το τελευταίο σχόλιο που είναι η καλή ποιότητα ζωής για τους πολίτες μας. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό που με ανησυχεί είναι το εξή. Σήμερα οι ασθενείς αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μία οδηγία σαν αυτή που έχουμε μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μικρό αριθμό ασθενών οι οποίοι γνωρίζουν πραγματικά τα δικαιώματα ε, τα οποία έχουν όταν λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη εκτός συνόρων. Πιστεύω πως αυτού του είδους τις δράσεις θα πρέπει να τις επεκτείνουμε σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανταλλάσσουμε, για παράδειγμα, βέλτιστες πρακτικές, το τι γίνεται σε μια χώρα και το τι γίνεται σε κάποια άλλη, έτσι ώστε να τα γνωρίζουν αυτά οι ασθενείς. Ένα δεύτερο που με απασχολεί. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, πολλές καθυστερήσεις Τη στιγμή λοιπόν της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων για την υγεία των ε, ασθενών, καθυστερήσεις μεταξύ χωρών, πώς μπορούμε αυτά να τα λύσουμε. Εγώ ζω στην άκρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον από εκεί προέρχομαι, και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον πώς λειτουργεί αυτή η ροή ασθενών, γιατί είναι τεράστιες οι διαφορές. Πολλές φορές δεν υπάρχει αρκετή συνεργασία μεταξύ ε, κρατών. Για παράδειγμα, με ασθενεί οι οποίοι φτάνουν από κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται στα, στις άκρες της επικράτειας. Κάτι που είπε μία συνάδελφος για τις σπάνιες ασθένειες. 26 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ασθενήσει από σπάνια ασθένεια και εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας οικονομικής δεν ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουμε αυτού του ασθενεί που ε, υποφέρουν από αυτέ τι σπάνιες ασθένειε. Είχατε πει ένα μηχανισμό χρηματοδότηση, πιο απλό, πιο διάφανο. Αυτή θα ήταν μια δυνατή λύση. Δεν ξέρω, είχετε κάποιε πληροφορίε παραπάνω να μου δώσετε γι' αυτό. Ήταν μια πρωτοβουλία. Θα ήθελα δηλαδή να μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτού που υποφέρουν από αυτές τις σπάνιες ασθένειες. Ε, Κύριε Welsh, Παρακαλώ, αν μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέρφων. Είσαστε επικεφαλής του νομικού τμήματος ε, Μάλλον όχι, θα ήθελα να παρακαλέσω τον επικεφαλής του νομικού τμήματος ε, της ε, Γενικής Διευθύνσης Σαντέ να πάρει το λόγο, αλλά ζητώ συγγνώμη, έχω άλλο ένα συνάδελφο που θέλει να πάρει το λόγο και κατόπιν θα σας δώσω το λόγο. Κυρία Χάζεκαμπ, ζητώ συγγνώμη. Α, όχι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, έχω μπερδευτεί. Μάλλον καλό θα είναι να εγκαταλείψω την Προεδρία πολύ σύντομα. Η κυρία Χάζεκάμ θα πάρει τη θέση μου. Αν λοιπόν να μας δείτε να, αλλάξουμε, αλλάζουμε θέσεις, αυτό ε, θα συμβαίνει. Πολύ ευχαριστώ. Ε, θα πάρω το λόγο πρώτος, διότι νομίζω ότι πολλές από τις ερωτήσεις αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει πρώτο το λόγο. Ωραία, θα κάνω ό,τι μπορώ με τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που ακούσαμε. Αρκετοί αναφέρθηκαν στο εξή. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε περισσότερα σχετικά με τι πραγματικέ ροέ των ασθενών σύμφωνα με την οδηγία και σύμφωνα με τον κανονισμό. Ε, πολύ θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα πάνω στο θέμα αυτό. Οι συνεργάτες μου και εγώ προσωπικά έχουμε εξετάσει επί αρκετό καιρό τις ροές αυτές. Προσπαθούμε να δούμε πού πηγαίνουν οι ασθενείς. Και προσπαθούμε να ε, κάνουμε περιστατωμένες υποθέσεις ε, σχετικά με το τι τους κινεί. Η Γαλλία έχει πολύ καλό σύστημα υγεία. Ε, δεν φαίνεται όλοι οι ασθενείς που φεύγουν από τη Γαλλία λοιπόν να, ζητούν καλύτερη περίθαλψη αλλού. Αυτό μπορεί να ισχύει για συγκεκριμένε ασθένειες, αλλά δεν φαίνεται αυτό αυτή να είναι η σημαντικότερη κινητήριος δύναμη. Η Γαλλία δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στους δύο μηχανισμούς, ε, της οδηγίας και του κανονισμού δηλαδή, από ό,τι γνωρίζω. Τα δύο τρίτα, τα εκατό δηλαδή των ασθενών ε, που ε, περνάνε τα σύνορα για περίθαλψη προέρχονται από ένα κράτος μέλος που δεν κάνει τη διάκριση ανάμεσα στους δύο μηχανισμούς και έτσι δυσκολεύονται οι ερευνές μας. Αρκετοί από εμά ζούμε σε κράτος μέλος ε, διαφορετικό από αυτό στο οποίο γεννηθήκαμε, οπότε είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουμε στην πατρίδα μα για περίθαλψη. Νομίζω ότι ε, σε μεγάλο βαθμό η διασυνοριακή περίθαλψη οφείλεται σε ανθρώπους Θα μπορούσε να φανταστεί κανείς δηλαδή από τα νούμερα ότι κάποιοι Εστονοί που εργάζονται στην ε, Φιλανδία παίρνουν την συνταγή του γιατρού από την ε, Φιλανδία αλλά την χρησιμοποιούν στην Εστονία. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Πρέπει όμως να εργαστούμε με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ίδιο. Η κυρία Μέρς νομίζω ότι έκανε μια πολύ σωστή παρατήρηση σχετικά με την πολυπλοκότητα του συστήματος για τους ασθενείς υπάρχουν περισσότεροι από έναν μηχανισμοί για επιστροφή των δαπανών. Ε, ζητώ συγγνώμη, μου φαίνεται ότι και εγώ χρειάζομαι τη συνολική περίθαλψη. Εν πάση έχουμε πολλές απαιτήσει από τους ασθενείς ε, όσον αφορά την κατανόηση των μηχανισμών αυτών. Εγώ προσωπικά μεσοπρόθεσμα θα ήθελα πολύ να εξεταστεί ο τρόπος απλοποίησης της οδηγίας αυτής, διότι νομίζω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Υπάρχει και το θέμα της ε, συνταξιοδότησης. Ε, βλέπουμε πολλές ε, μετακινήσεις ανθρώπων από τις κρύες χώρες στις πιο ζεστές. Όσον αφορά την χρήση των συστημάτων πληροφορικής, υπάρχει ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τη Γενική Διεύθυνση Υγείας, την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ, αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση των προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με συστήματα πληροφορικής. Θα πρέπει να έχουμε ε, πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το πόσο θα στοιχήσουν και το τι αποτέλεσμα θα επιφέρουν. Τα ίδια τα κράτη-μέλη μπορεί να έχουν πολύπλοκα συστήματα υγείας και γι' αυτό ακόμη και ε, σε εσωτερικό επίπεδο μας ενδιαφέρουν οι ανταλλαγές δεδομένων με βάση την ηλεκτρονική υγεία, το e-health. Επίσης, το ότι σχεδιάζεται ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε δύο κράτη-μέλη δεν σημαίνει ότι ο κάθε πάροχος υπηρεσιών υγείας ε, θα πρέπει να στέλνει δεδομένα σε άλλη χώρα. Μπορεί αυτό να ισχύει για περιορισμό αριθμό ε, φορέων. Ενώ προχωρούν οι εργασίες μας, αναρωτιέμαι εάν Αναρωτιέμαι κατά πόσο θεωρείται σύγχρονο το σύστημα αυτό. Μπορεί να φαινόταν σύγχρονο πριν 10 χρόνια, αλλά σήμερα δεν είμαι βέβαιος ότι είναι πια κατάλληλο και δεν έχω κάποια λύση να σας προτείνω. Δεν νομίζω ότι η απάντηση στην περιορισμένη επιτυχία που έχουμε σε κάποια από τα θέματα αυτά είναι να δαπανίσουμε περισσότερο χρόνο. Πιθανότητα να πρέπει να εξετάσουμε αν υπάρχει άλλος τρόπος να λύσουμε ε, το συγκεκριμένο πρόβλημα. Νομίζω ότι απάντησα έτσι στις ερωτήσεις ε, που θεωρώ ότι μπορώ να απαντήσω. Πολύ ευχαριστώ. θα επανέλθω με πρόσθετες πληροφορίες. Θα προτιμούσα πάντως ε, να επανέλθω αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλάβει τα καθήκοντά της και μας δώσει στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα. παρακαλώ, το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ το Ενακτικό Συνέδριο που μας βοηθά ιδιαίτερα στη δουλειά μας. Η υγεία είναι εθνική αρμοδιότητα, μην το ξεχνάμε. Και έτσι και στις ανταλλαγές των στοιχείων για τον ασθενή αλλά και στην ανάπτυξη ε, των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο μπορεί να επηρεάσουν ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση αυτών των ανταλλαγών αλλά και την ανάπτυξη των δικτύων. Τα εθνικά συστήματα. Ευχαριστούμε λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο. Οι παρατηρήσεις του θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε περαιτέρω την οδηγία για την ίδια την οδηγία έχουμε δύο νομικά πλαίσια τον κανονισμό και την οδηγία προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε σημεία επαφής για την οδηγία ώστε να συνδυάζονται τα δύο αυτά κείμενα Το πρώτο ορίζει τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η αγωγή σε εξωτερικό και το άλλο είναι η παροχή υποστήριξη και η βοήθεια σε κάποιον που είναι κατεστημένος στο εξωτερικό. Όλα αυτά έχουν να κάνουν λοιπόν με την υλοποίηση της οδηγίας. Δύο εκατομμύρια χρήστες της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης έχουν ωφεληθεί από τον κανονισμό λιγότεροι ε, είναι αυτοί που μπορεί να έχουν ωφεληθεί από την οδηγία, αλλά ίσως η εξέλιξη αυτή να είναι και φυσιολογική και προσπαθούμε να ενισχύσουμε την υποστήριξη από τα εθνικά σημεία υποστήριξης. Έχουμε ενισχύσει το εργαλειοθήκη και έχουμε δώσει τα απαραίτητα στοιχεία. Για τις δομές πρέπει να επενθυμίσω από την αρχή ότι είναι μια διαδικασία καινούργια για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αρχών, στηρίζεται σε θελοντική βάση, 22 κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ανταλλαγές ως το 2022, σταδιακά. Υπολογίζουμε ότι τα υπόλοιπα ως το 2027 θα έχουν και αυτά ενταχθεί. ώστε να έχουμε και τα εθνικά σημεία επαφής με την υποστήριξη βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ταμείο Συνδέοντας στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη βέβαια θα εξαρτηθεί πολύ, η ανάπτυξη των υποδομών, από το ε, εθνικό επίπεδο. Κάποια κράτη-μέλη πρόσφατα εισήγαγαν την νομοθεσία και ζητούν ε, ηλεκτρονικά μητρώα υγείας ε, και άρα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική ένα κράτος μέλος παρακολουθούμε σε βάση τριμηνία Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου είχαμε πληροφορίες από τη Φιλανδία κυρίως και την Εστονία, με 2.700 ηλεκτρονικές συνταγές ε, για Ευρωπαίους πολίτες στην Εστονία ήδη. Διμερώς βλέπουμε ότι έχουν φτάσει στις 4.000 συνταγές, 30 Τσεχική Δημοκρατία και Κροατία με την ε, ανταλλαγή ηλεκτρονικών σταγών και πάλι περιμένουμε να έχουμε περισσότερη ενημέρωση σύντομα. Η Μάλτα και η Πορτογαλία έχουν επίσης λάβει το σχετικό πράσινο φως για τις ανταλλαγές. Και έτσι παίρνουν πια στην υλοποίηση αυτό που ονομάζουμε φάση παραγωγής εμείς. και περιμένουμε την ενημέρωση τον επόμενο μήνα. Η κατάσταση έχει να κάνει βέβαια και με τη διαλειτουργικότητα που είναι κάπως άνηση. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη στην ανταλλαγή αυτών των ηλεκτρονικών μητρών. Έχουμε τη σχετική σύσταση για τις προδιαγραφές, τα τεχνικά, τεχνικά στοιχεία, τους όρους που θα εξασφαλίσουν την ανταλλαγή αυτή κατά τρόπο ασφαλή. Όταν υλοποιηθεί αυτό πιστεύουμε ότι θα δούμε και μια ενίσχυση στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών μητρών, ίσως ηλεκτρονικών ιστορικών, ίσως όχι μεταξύ όλων των κρατών αλλά τουλάχιστον μεταξύ όμορων. Ανταλλαγή πληροφοριών που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε εξοικονόμηση πόρων, γιατί θα χρειάζονται να επαναληφθούν κάποιες ε, εξετάσεις εργαστηριακές αναλύσεις, ε, τομογραφικές αναλύσεις κτλ. Και για το ERN που είναι ένα σχέδιο πολύπλοκο πάνω από 300 ε, νοσοκομεία έχουν ενταχθεί στα δίκτυα αυτά. Έχουμε διάφορους συμβεβλημένους εταίρους επιπλέον νοσοκομεία που αποτελούν ε, σημείο αναφοράς για τους ασθενείς που έχουν ε, σπάνιες ασθένειες. Έχουμε πάνω από 200, 200 φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας στα κράτη-μέλη. Τις επόμενες εβδομάδες ε, γίνεται προκήρυξη και για, για νέα μέλη. Ωστόσο, πρόκειται και μια διαδικασία στην οποία χρειαζόμαστε υποστήριξη από τα κράτη. Εμείς προσφέρουμε ένα εργαλείο που επιτρέπει την ε, συζήτηση, την επικοινωνία για σπάνιες ασθένειες και έτσι έχουν αναπτυχθεί 740 πάνελ συζήτησης. Πάνω από 2.000 είναι γιατροί που έχουν συνδεθεί στο σύστημα και ανταλλάσσουν πληροφορίες Προσπαθούμε σε συνεργασία μαζί τους να κάνουμε πιο ευέλικτο και ταχύ το σύστημα και να το προσαρμόσουμε σε ανάγκες τους. Προσπαθούμε να το συνδυάσουμε ώστε να υποστηρίξουμε και ε, τις, τα εθνικά συστήματα. Υποστηρίζουμε τα δίκτυα και στην επιτήρηση, στην παρακολούθηση των ε, δράσεων, πράγμα το οποίο θα αργήσει να δώσει αποτελέσματα. Η αξιολόγηση τους θα γίνει το 2020-2023. Υποστηρίζουμε την έρευνα και ανάπτυξη, σημαντικά κομμάτια των δικτύων που προσφέρουν την προσθέμενη αυτή αξία για τις σπάνιες ασθένειες στην Ευρώπη. Όλα αυτά βέβαια είναι απλά και θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω το ρόλο των ε, κρατών, αλλά και το δικό σας που μπορείτε να υποστηρίξετε αυτές τις προσπάθειες με τη χρηματοδότηση. Έχουμε από το Ταμείο την ε, σχετική υποστήριξη, έχουμε τη διοικητική υποστήριξη, έχουμε ένα εκατομμύριο ευρώ ανά, έτος, 200 ε, ανά πενταετία, 200.000 το έτος και Υποστηρίζουμε έτσι τα κράτη που στηρίζουν τους συντονιστές σε εθνικό επίπεδο Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο ιδιαίτερως έχουν ξεκινήσει συστηματική αυτή την προσπάθεια ευπρόσδεκτη προσπάθεια και για τους συντονιστές αλλά και για τους ε, ασθενείς και τις οργανώσεις ασθενών. Το πολιετές νοσονομικό πλαίσιο προβλέπει στο τμήμα που αφορά την ψηφιακή Ευρώπη υποστήριξη και με το Ταμείο βέβαια συνδέοντας την Ευρώπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε να κατηδρήσουμε αυτό το σύστημα πληροφορικής αλλά και σε επίπεδο συντονιστών ε, θηρίδες για τα νοσοκομεία, ένα νέο σχέδιο καινοτόμο, χρήσιμο, η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, οι συντονιστέ και εσείς με τα βήματα που αναλαμβάνετε, προχωράτε βήμα-βήμα για τη βελτίωση των παρεχομένων στον ασθενή υπηρεσιών. Είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Είναι πολλέ οι προκλήσει βέβαια που έχουμε μπροστά μα και δεν μπορούμε εμεί να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Στο επίπεδο τη Επιτροπή χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων και του καθενός και ελπίζω η εκθέση του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά και η δική σας υποστήριξη να, μας, ε, να αποδειχθούν χρήσιμες και στις δικές μας προσπάθειες. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάω δεξιά αριστερά. Έχουμε άλλα μέλη που να θέλουν κάτι να ρωτήσουν. Παρακαλώ. Έχει μείνει κάτι αναπάντητο. Βλέπω έναν τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς για την παρουσίασή σας και θα ήθελα και να σας συγχαρώ για την θετική σας εμπλοκή έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη κινητικότητα για τους ασθενείς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ πως τα η διασυνοριακή περίθαλψη δίνει ευκαιρία στους Ευρωπαίους πολίτες για να ε, ψάξουν πού είναι η καλύτερη ιατρική περίθαλψη για την περίπτωσή τους και σε μερικό πλήρως να αποζημιωθούν για αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι ένα από τα πολύ θετικά επιτεύγματα των περασμένων ετών στον κλάδο της υγείας και είναι καλό να έχουμε αυτή την άριστη εφαρμογή της οδηγίας. Δύο είναι τα μεγάλα εμπόρια, ε, ε, εμπόδια με τα οποία δεν επιτρέπουν στους ασθενείς να αναζητήσουν περίθαλψη σε άλλο ε, κράτος μέλος από αυτό της καταγωγής. Καταρχήν, ποια είναι η δυνατότητα αποζημίωσης αυτών των δαπανών και τι συμβαίνει σε κράτη-μέλη άλλα. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό υγείας του κράτους μέλους. Ήμουνα για ένα χρόνο επικεφαλής του Εθνικού Ασφαλιστικού Οργανισμού Υγείας ε, στη Ρουμανία και πραγματικά το όριο για την αποζημίωση ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Εκτός λοιπόν από τις πιέσεις του προπολογισμού υπάρχουν και προβλήματα γραφειοκρατικά ή διαδικασιών σε κάποια κράτη-μέλη που δυσκολεύουν πάρα πολύ την κατάσταση και αρκετοί ασθενείς αποθαρρύνονται και δεν ζητούν να τους καταβληθεί η αποζημίωση για τις δαπάνες που έχουν κάνει, κυρίως όταν είναι μικροποσά. Επίσης, η προτεραιότητα που δίδεται και εδώ χρειάζεται μια συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης έτσι ώστε να δούμε σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται προέγκριση και γιατί καμιά φορά ζητάνε προέγκριση χωρίς να υπάρχει λόγος. Επίσης, είναι επιτυχημένο το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφορών, είναι σημαντική εξέλιξη του e-health με την ηλεκτρονική διασύνδεση και είναι σημαντική διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων μας. Γιατί όταν αντιμετωπίζουμε μια περίπτωση όπου ε, μπορούμε να μεταφέρουμε μέσω διασυνδεσιμότητας τα, ε, το φάκελο του ασθενή από τη μία χώρα στην άλλη, τότε η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αυξάνεται. Και κυρίως για τους ασθενείς οι οποίοι αναζητούν περίθαλψη και ιατρική φροντίδα σε παραπάνω από ένα κράτη-μέλη. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι. Νομίζω πως η δήλωσή σας σε κάποιο βαθμό έχει ήδη απαντηθεί. Δεν ξέρω αν οι ομιλητές θέλουν κάτι παραπάνω. Για τη στήριξη που προσφέρουμε στα κράτη-μέλη για το σύστημα επιστροφών και αποζημιώσεων, αυτό που κάνουμε τώρα είναι ο διμερής διάλογος και οι βέλτιστες πρακτικές και σεμινάρια σχετικά. Και στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η οδηγία, τότε η διαδικασία επιπαραβάσει. Άκουσα μια σειρά παρεμβάσεις για τα ορφανά φάρμακα. Αυτό βεβαίως δεν καλύπτεται από την οδηγία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αξιολογεί αυτή τη στιγμή τη σχετική νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Μια τελευταία παρατήρηση. Πολύ σύντομες ερωτήσεις. Ρωτώ. Για το δίκτυο αναφοράς, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε σύσταση ισχύρη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στα επίσημα στα εθνικά συστήματα υγείας. Και τότε έχουμε και τη βιωσιμότητα και τη χρηματοδότηση και όλα. Και σε εσάς, ελεκτικό συνέδριο, ρωτώ το εξή. Αν αναλύσετε τα υπέρ και τα κατά αυτή τη διαδικασία προέγκριση. Γιατί υπάρχουν επιχειρήματα και υπέρ. Και σας ρωτώ μάλλον, το εξετάσατε το σύστημα της προέγκρισης, γιατί ίσως ε, σε κάποιο βαθμό περιορίζει ε, την μετακίνηση μέσα στην Ευρώπη. Οπότε πείτε μου, έχετε κάνει οτιδήποτε σχετικό. Στα γρήγορα λοιπόν να μας απαντήσετε. Καταρχήν το αμέλησα. Δεν μίλησα για τις βέλτιστες πρακτικές, για την παροχή υπηρεσιών. Η ομάδα μου μου λέει ότι μάλλον η Σουηδία ήταν η καλύτερη στο βαθμό στον οποίο ενημερώνει τους ασθενείς και κυρίως ενημερώνοντάς τους για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Συμφωνώ. Υπάρχουν πολλά θέματα για τον τρόπο που αποζημιώνεσαι για τις δαπάνες στα διάφορα κράτη-μέλη. Ειλικρινά δεν βλέπω πώς μπορούμε να το παρακάμψουμε, γιατί είναι εθνική αρμοδιότητα η ιατρική περίθαλψη. Και ο καθένας οργανώνει το δικό του εθνικό σύστημα υγείας με διαφορετικό τρόπο. Πάντα θα υπάρχουν αυτές οι δισκαμψίες στα σύνορα. Έχουμε σκεφτεί πολύ το πόσα κράτη-μέλη έχουν εθνική στρατηγική για τις ε, σπάνιες και σε πόσες από αυτές έχουμε ένα βαθμό διασυνοριακής συνεργασίας. Ίσως λοιπόν έχουμε περιθώριο μέσα στις ίδιες εθνικές πολιτικές, αλλά δεν έχω νομίζω να πω. Δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι θέλουν να απαντήσουν. Um, Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, μπορούμε να το κλείσουμε το σημείο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα για εμάς. Και θα τα ξαναπούμε στο μέλλον, σίγουρα. Πριν κλείσω τη συνεδρίαση να σας πω πως θα ξεκινήσουμε στις 2.30 με την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Βέλα για τη βιοπικιλότητα. Άρα λοιπόν σας εύχομαι καλή όρεξη και θα τα πούμε το απόγευμα.